Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ήδη καθυστερήσει λίγο και έχουμε πολύ περιφορτωμένο πρωινό πρόγραμμα και περιορισμένο χρόνο, γιατί όπως σας είπα, στα 10 παρατέταρτο θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, μια και οι συντονιστές θα συναντήσουν τον Υφυπουργό Γουατλέ και κλεισμένο των θυρών. Περιμένοντας να καθίσετε και να προετοιμαστείτε για τις ψηφοφορίες, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο που φέρνει τους Γάλλους να εργάζονται στις 14 Ιουλίου. Ε, εθνική εορτή, η μέρα της Βαστίλης. Για να φανταστείτε τι πολιτικό βάρος έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναγκάζει τους Γάλλους να εργάζονται τέτοια μέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γραμματεία, τη, τους συνεργάτες ε, της ομάδας για τις άοκνες προσπάθειές τους προκειμένου να προετοιμάσουν τη σημερινή ψηφοφορία. Και ξέρω ότι οι πόρτες του Μιγγέλ Πόρτας έμειναν διάπλατα νυχτές όλο το βράδυ για να συνομιλήσει με τους ενδιαφερόμενους για τις συμβαστικές λύσεις. Έχουν αναθεωρηθεί μερικές συμβαστικές λύσεις. Σας έχουν ε, αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η συμβαστική λύση ΚΑΠΑ για την παράγραφο 9 και η συμβαστική λύση ΔΕΛΤΑ στην αιτιολογική σκέψη ΕΛ, που είναι μια φιλοσοφική συμβαστική πρόταση που έκανε ο κύριος Μπογκρός για το χαρακτηρισμό της παγκοσμιοποίησης. Έχετε λάβει όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας και τις δύο νέες συμβαστικές προτάσεις. τη σελίδα με τις δύο συμβαστικές προτάσεις, Κ και Δ. Ο κύριος Άγκλουντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι οι φιλελεύθεροι θέλουν ψηφοφορία κατά τμήματα για το Κ, παρόλο που αναδιατυπώθηκε η συμβαστική λύση. Δεν αναφέρεται στον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά ευελπιστούμε ότι θα μας επιτρέψετε να ψηφίσουμε κατά τμήματα. Καλά, θα το δούμε όταν ψηφίσουμε το ΚΑΠΑ. από εκεί που λέει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση της ε, περίπτωσης ε, ίδρυσης ξεχωριστού ανεξάρτητου ταμείου. Από εκεί και πέρα θέλουμε ξεχωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα, όπως είχαμε πει και πριν την αρχική συμβαστική πρόταση. Καλώς, το σημειώνουμε. Άλλες παρατηρήσεις για τις ψηφοφορίες υπάρχουν. Ευχαριστώ. Περνάμε στην έκθεση, ψηφοφορία έκθεση πόρτα. Για την παράγραφο 1... Μία διευκρίνηση. Και εγώ μπορώ να ψηφίσω, γιατί δεν έχει απαρτία το ΑΕΛΚ. Για την συμβαστική λύση ε. Ποιος είναι υπέρ της συμβαστικής λύσης ε του εισηγητού. Κατά. Κατά, κατά της συμβαστικής πρότασης ε. Αποχές. Ωραία, ευχαριστώ, εγκρίνεται. Οπότε οι τροπολογίες 22 με 25... Όχι, μάλλον 22 και 23 μόνο καταπίπτουν. Συμβαστική λύση F του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική λύση G. G. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική λύση H, ψηφοφορία κατά τμήματα, αναφέρεται στο φύλλο της ψηφοφορίας. Πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, πρώτο τμήμα του H, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ποιος είναι υπέρ, κατά Αποχές. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική λύση ή Ποιος, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή εγκρίνεται και συμβαστική λύση Συμβαστική λύση η συμβαστική λύση I καλύπτει τις τροπολογίες 43, 44 και 45, αλλά δεν καλύπτει 46, οπότε θα ψηφίσουμε την τροπολογία 46 του κύριο Άλβαρο και λοιπόν αφιλελευθέρων, Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Καταμέτρηση αλλά νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία παρόλα αυτά. Ποιος είναι υπέρ και πάλι για να μετρήσουμε. κατά αποχές σαφής πλειοψηφία διακρίνεται υπέρ του 46 47, ο εισηγητής είναι κατά γι' αυτό υπέρ, ποιος είναι υπέρ της 47 κατά αποχές το 47 απορρίπτεται η 48 καλύπτεται τροπολογία 49 τώρα του ΕΛΚ ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία J. Το ΕΛΚ ζήτησε ψηφοφορία κατά τμήματα. Ο κύριος Χάγκλουντ. Κύριε Πρόεδρε, θεωρούμε ότι η τροπολογία 55, παρόλο που αναφέρεται ότι καλύπτεται, κατά τη γνώμη μα ε, δεν καλύπτεται, γιατί θα θέλαμε να την ψηφίσουμε ξεχωριστά και δεν εμπίπτει στη συμβαστική τροπολογία J. Ωραία. Την 55 ξεχωριστά. Θεωρείτε ότι δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία J, έτσι. Θα την ψηφίσουμε μετά. Προ το παρόν για τη συμβαστική τροπολογία J. Πρώτο τμήμα. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο άλλο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Το πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. ίδια πλειοψηφία με πριν. Αποχές. Η υπέρ. Εγκρίνονται και τα δύο τμήματα της συμβαστικής τροπολογίας. Α, λάθος λέει πρώτα. Συγγνώμη. Ε, δεν πρόλαβα να πιω καφέ. Δεν ξέρω αν εσείς πιέτε, πάντως εγώ δεν είδα καφέ προς το παρόν. Ωραία. Το δεύτερο τμήμα απορρίπτεται. Καλύφθηκαν οι τροπολογίε σε 50, 54, 51, 52 και 53. Και πάμε στην 55. Νομίζαμε ότι καλυπτόταν από την τροπολογία της συμβαστική J, αλλά οι φιλελεύθεροι διαφωνούν και ζητούν ξεχωριστή ψηφοφορία για την τροπολογία 55. Ο συγκητής τι γνώμη έχει. Είναι κατά. Καλώς. Δέχομαι να ψηφίσουμε ξεχωριστά την τροπολογία 55. Κατά τη γνώμη μου όμω η διατύπωση τη συμβαστικής τροπολογίας J λέει το ίδιο πράγμα και μάλιστα σαφέστερα. Εγώ σας προτείνω να ψηφίσετε κατά γιατί κατά τη γνώμη μου το περιεχόμενό της καλύπτεται αλλά αξιοσέβαστη η γνώμη των φιλελευθέρων. Καλώς, ακούσατε τώρα εισηγητή. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 55. Κατά. Αποχές. Η τροπολογία 55 απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία K. Αναθεωρημένη. Ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα. Κύριε Χάγκλουντ, ζητήσατε να διαχωρίσετε το τμήμα που λέει ότι θεωρείται ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξέταση της πιθανότητας ίδρυσης ανεξάρτητου ταμείου με ξεχωριστές δεσμεύσεις, ε, υποχρεω... Ε, υποσχε... και πληρωμών μέχρι το τέτοιο ταμείο. Αυτό ξεχωριστά. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Και το τρίτο. Ποιος είναι υπέρ. Με εξαίρεση λέει, το, το τμήμα που πρότεινε φιλελεύθερη. Κατά. Αποχές. Χωρίς αποχές. Οπότε το πρώτο τμήμα και το τέλος, από εκεί που λέει ε, θεωρεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση και το πρώτο τμήμα μέχρι το εξετάζει ε, Ποιος είναι υπέρ τώρα του δεύτερου τμήματο. Θεωρεί ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και τα λοιπά. Μέχρι το τέτοιο ταμείο. Ποιο είναι υπέρ. Δεν θέλω να εμπλακώ στα εσωτερικά του ΕΛΚ, αλλά κανονικά το ΕΛΚ θα πρέπει να είναι υπέρ, αφού ήταν υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας. Δεν ξέρω, εντάξει, εσείς θα κανονίσετε. Ποιος είναι υπέρ, υπέρ Μπάρμπαρα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, μήπω μπορούμε να επαναλάβουμε αυτή την ψηφοφορία, γιατί νομίζω ότι και εγώ δεν τα κατάλαβα καλά, γιατί και εγώ δεν έχω πιει καφέ σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. donc, Αν κατάλαβα καλά, οι φιλελεύθεροι ενοχλήθηκαν από την ενδιάμεση πρόταση και θέλουν ξεχωριστή ψηφοφορία για να εκδηλώσουν τη διαφωνία τους με τη φράση αυτή. Εγώ κατάλαβα ότι οι υπόλοιπε ομάδε συμφωνούν με ολόκληρη τη συμβαστική τροπολογία ΚΑΠΑ. Οπότε είναι λογικό οι υπόλοιπε ομάδε να υπερψηφίσουν ολόκληρη τη συμβαστική τροπολογία ΚΑΠΑ. Εκτό και αν η αφαίρεση αυτή τη φράση του ενοχλεί. Καταλάβατε, κυρία Βαρβάρα. Μάλιστα. Για το δεύτερο τώρα τμήμα. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ. Και η κυρία Βαρβάρα είναι υπέρ. Και οι υπόλοιποι βουλευτέ είναι υπέρ. Όλοι υπέρ. Κατά. Κατά οι φιλελεύθεροι. Το είχαν δηλώσει από την αρχή. η πρασινη επίση είναι κατά και κάποιοι άλλοι. Αποχέ. Θαυμάσια. Πάντω πλειοψηφία υπάρχει υπέρ τη διατήρηση τη φράση αυτή και τη διαφύλαξη ολόκληρη συμβαστική τροπολογία ΚΑΠΑ. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία L. Και εδώ ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα. Ο εισηγητή είναι υπέρ και των δύο τμήματων. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματο. Πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Για το πρώτο τμήμα, ποιο είναι υπέρ. Κατά. Je remercie. Abstention. Αποχές. Εγκρίνεται με μικρή διαφορά υπέρ για το πρώτο τμήμα τώρα. Δεύτερο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 67 του κυρίου Μάνερ που δεν καλύπτεται. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ είναι η φιλελεύθερη κυρία Ανδρέασεν. Κατά ποιος είναι η πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται, αποχές. Πέντε αποχές. Απορρίπτεται. Η 68 καλύπτεται. Η 69 όχι. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70. Πανομοιότυπη με την 69. 71. Ε, ζητά συγγνώμη που αποουσιάζει η κυρία Βέρτμαν. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πλειοψηφία. Αποχές. Μία αποχή. Άρα απορρίπτεται η τροπολογία 71. Τώρα για τις αιτιολογικές σκέψεις. Συμβαστική τροπολογία α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ωραία, εγκρίνεται. Δεν καλύπτει όμως την τροπολογία 3 του ΕΛΚ. Ποιος είναι υπέρ. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Κατά. Abstention. Αποχές. Il est adopté par une légère... Με ελαφρά διαφορά, με ελαφρά πλειοψηφία εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Ο εισηγητής είναι υπέρ, φυσικά δική του είναι. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, χωρίς αποχές, εγκρίνεται. Δυστυχώ δεν καλύπτει και πολλέ άλλε τροπολογίε, οπότε θα ψηφίσουμε τι τροπολογίε χωριστά. 7. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 7. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Ο εισηγητή είναι κατά. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, ε, δεν δικαιούμαι πια να ψηφίζω. Δεν ψήφισα και πολύ τόσο άλλο, σε πάση περιπτώσει. Τροπολογία 9 ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Λαβία. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. κατά αποχές τα δύο άκρα είναι υπέρ εγκρίνεται πολύ διασκεδαστική αυτή η αλλαγή των ε, πλειοψηφιών βλέπω ότι περάσατε πραγματικά πολύ δύσκολη νύχτα και εργαστήκατε πραγματικά όκνα για το 11 καταπίπτει 9 ε, ναι, συγγνώμη η 10 έχει εγκριθεί η 11 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία C. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται. Καλύπτει τις τροπολογίες 12 και 13, αλλά δυστυχώς όχι και τη 14. Ψηφίζουμε τη 14. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ε, αποχές η αριστερά είναι μια ψηφία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ο εισηγητής είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ο εισηγητής είναι υπέρ τελικά. Καλά. Άνθρωπος. Δικαιούται να αλλάξει γνώμη. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Γιατί 15. Εγκρίνεται. Τελικά δεν καταλάβαμε. Ήταν υπέρ ή κατά ο εισηγητής. Ναι. Θα μείνει άγνωστο. Αναθεωρημένη συμβαστική τροπολογία Δέλτα. Ποιο είναι υπέρ. Ντε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δύο τροπολογίες έχουμε που δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές ε, τροπολογίες. Το 20, ο εισηγητής είναι κατά του, της κυρίας Μάνερ. Ποιος είναι υπέρ. Συγγνώμη κυρία Μάνερ που σας είπα κύριο. Αλλά Μάνερ, όνομα είναι αυτό για γυναίκα, είναι περίεργο λίγο. Ανδροπούλου. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ιτήθηκε η κυρία Μάνερ. Απορρίπτεται την τροπολογία της. Τελευταία τροπολογία Βέρτμαν 21. Ο εισηγητής είναι κατά. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά. Αποχές χωρίς αποχές, οπότε απορρίπτεται. Θα ψηφίσουμε τώρα μαζί τις δύο γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών και Απασχόλησης. Θα ψηφίσουμε από κοινού τις διατροπολογίες για να, δούμε, να πούμε τι καλύπτονται. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ των δύο γνωμοδοτήσεων για να αποτίσουμε στις δύο επιτροπές που έδωσαν τις γνωμοδοτήσεις και να δείξουμε ότι τις λάβαμε υπόψη. Κατά αποχές, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Σας ευχαριστώ. Τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να μετρήσουμε. Καλύτερα για τα πρακτικά. Και πάλι, ποιος είναι υπέρ στην τελική ψηφοφορία. Εγώ δεν ψηφίζω. Κατά. 30 ήταν υπέρ. Εννέα κατά. Αποχές. Μία αποχή. Οπότε εγκρίθηκε η έκθεση. Χαρητήρια κύριε Σιγητά. Ήταν πραγματικά αξιέπαινο το έργο σας και το δικό σας και των συντονιστών. Πολύ αξιόλογο. Γιατί συμβάλλατε όλοι στην διαμόρφωση των συμβαστικών τροπολογιών. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία για την έκθεση Γκάιερ. Voilà, simplement, le président aurait besoin de la liste de vote. Ναι, αν μπορούσε κάποιος να μου δώσει τον κατάλογο ψηφοφορίας. Voilà. Alors, alors j'ai plusieurs demandes de parole έχω κάποια αιτήματα λόγου. Πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο εισηγητής νομίζω πως θέλει να πάρει το λόγο και επίσης ο κύριος Λαβία και ο κύριος Άγγλουντ μου ζήτησαν να πάρουν το λόγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Κύριε Γκάιερ, κύριε εισηγητά, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σύντομα βεβαίως, πρόκειται για γνωμοδότηση της Επιτροπής μας επί που κάνει η Επιτροπή Ήτρε που έχει λάβει ως αφορμή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπει 114 εκατομμύρια ευρώ πόρων που δεν έχουν διατεθεί να διατεθούν για μια χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων ενεργείας. Εμείς έχουμε προτείνει ορισμένες τροπολογίες. Με την ευκαιρία ευχαριστώ τις συναδέλφους και τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που επίσης κατέθεσαν τροπολογίες, τις οποίες μάλιστα δέχομαι όλες. Μάλιστα, αν δεν έχει κανείς ένσταση, μπορούμε να τις ψηφίσουμε και όλες μαζί, ευθύς αμέσως. Διότι και από την άλλη πλευρά έχω λάβει μηνύματα θετικά σχετικά με τις τροπολογίες. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις. Κάποια προβλήματα έχουμε από άποψη δημοσιονομικής τεχνικής σχετικά με 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία βρίσκονται στον τίτλο 2 και τα οποία υποτίθεται θα προσθεθούν στα 114 εκατομμύρια. Την ιδέα αυτή είχε η κυρία Βαν Μπρέμπτ της Επιτροπής Ήτρε. Και εγώ συμφώνησα. Αυτά τα 15 εκατομμύρια δεν έχουν νομική βάση για να είναι στην, στον τίτλο 2 και αν δεν τα διαθέσουμε διαφορετικά θα χαθούν. Με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό το συζητήσαμε τεχνικά Εάν υπάρχει παρόν εκπρόσωπος της Κομισιόν θα ήθελα να τοποθετηθεί για να δω πώς το βλέπει αυτό το πράγμα. Εάν δηλαδή τα 15 εκατομμύρια θα πρέπει να παραμείνουν εκεί όπου είναι, δηλαδή στο τίτλο 2 χωρίς νομική βάση ή αν πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Αν μπορεί να συμφωνήσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την μεθοδολογία μεταφοράς. Νομίζω ότι θα αρκεστώ σε αυτά τα εισαγωγικά λόγια. Ευχαριστώ και πάλι για την συνεργασία και αναμένω την ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ. Ελαβία. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει μια απάντηση όσον αφορά αυτό το θέμα των 15 εκατομμυρίων. Γιατί ε, καταρχήν εγώ ε, δεν συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν ε, χρήματα του Leading 2 σαν να ήταν πιστοτική κάρτα έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν μέτρα άλλων παρεμβάσεων που δεν έχουν καμία σχέση με, την, με τις γεωργικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι συμβαίνει γιατί διαφορετικά εγώ θα καταψηφίσω, θα καταψηφίσω την ε, τροπολογία. Πρόεδρος, καταλαβαίνω κύριε Λαβία, από αυτά που μου λέτε ότι υπό την αίρεση της απάντησης της Επιτροπής θα καταψηφίσετε την τροπολογία 8. Δηλαδή, εάν έχετε ένα πρόβλημα, αυτό είναι το, η τροπολογία 8, γιατί ο εισηγητή πρότεινε να ψηφιστούν αμπλόκ οι τροπολογίες, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σα, εάν η απάντηση που θα λάβετε για την τροπολογία 8 δεν είναι σαφή, τότε εσεί θα καταψηφίσετε την τροπολογία 8. Πολύ ωραία. Επόμενος ομιλήτη, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω το ίδιο πρόβλημα με τον κύριο Λαβία. Γι' αυτό λοιπόν αναμένω και εγώ την απάντηση. Αλλά θα ήθελα να κάνω και μία ε, παρατήρηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Ξέρετε, είχαμε μονάχα 10 ώρες πριν να εκμεύσει η ε, προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών και παρακαλούμε για μία ακόμα φορά την γραμματεία να μας δώσει λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν είναι δυνατόν, είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση μέσα σε 10 ώρες να πρέπει να υποβάλουμε με τροπολογίες. Ε, δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά. Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο και με απασχολεί λίγο το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και έχετε δίκιο ότι δεν είναι παραδεκτές, δεν είναι σωστές ε, ε, ε, ε, συνθήκες εργασίας. Και πρέπει να σας πω όμως ότι δεν ευθύνεται η γραμματεία, ευθύνομαι εγώ γιατί αποφασίσαμε στους συντονιστές να πάρουμε έτσι να κάνουμε αυτήν την να δώσουμε αυτή την προθεσμία επομένως εγώ είμαι ο μόνος ναι, το πρόβλημα είναι η τροπολογία 5. Είναι η τροπολογία 5, λέει ο κύριος Λαβία. Έκανα λάθος προηγουμένως. 5-5 έχει δίκιο ο συνάδελφος. Είναι η τροπολογία 5, μπερδεύτηκα. Ωραία. Η κυρία Καρβάγιο. Ευχαριστώ πολύ. Ως σκιώδης συγγήτρια από το ΕΛΚΑ πρέπει να πω ότι στηρίζουμε τον εισηγητή και την χρήση των 15 εκατομμυρίων ε, το ΧΕΔΙ ε, αλλά ε, μονάχα για δράσεις που θα αφορούν την κλιματική αλλαγή. Ε, τώρα, όσον αφορά αυτούς που δεν συμφωνούν με την χρήση χρημάτων της επικεφαλίδας 2 που όντως αφορά γεωργικά θέματα, τι να σας πω μπορούν να ε, καταψηφίσουν την τροπολογία αυτή. Εμείς, επομένως, προτείνουμε on block τροπολογία, ε, ψηφοφορία εκτός από την τροπολογία 8, λέει η κυρία Καρβάγιο. Και όσοι θέλουν, όσοι δεν συμφωνούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά έτσι ώστε να δημιουργηθούν ε, ενεργειακά επαρκή κτίρια, τότε να καταψηφίσουν την τροπολογία αυτή. Επομένως, λέει ο Πρόεδρος, ε, υπάρχει και πειθαρχία και δημοκρατία ε, και ελευθερία ψήφου στο ΕΛΚ από ό,τι καταλαβαίνουμε. Άψογα. Βλέπω όμως ότι η Αν Γένσερ έτσι κουνάει το κεφάλι της με σκεπτικισμό στην παρατηρήσή μου, δεν έχει σημασία. Θέλετε το λόγο κύριε Ισηγητά, παρακαλώ. Ναι, ναι, πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να διευκρινίσω και πάλι ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε σημαντικές ανατροπές της μεθοδολογίας εργασίας της Επιτροπής μας. Πρόκειται για μια μεταφορά και παρακαλούμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πρόταση τεχνικής προσαρμογής. Περί αυτού πρόκειται. Τα ανώτατα όρια στις διάφορες κατηγορίες του προϋπολογισμού πρέπει να προσαρμοστούν. Αυτό είναι όλο. Έχω κατανόηση εάν για λόγους συστημικούς ορισμένοι συνάδελφοι του Λαϊκού Κόμματος μπορεί να διαφωνούν με την τροπολογία μου υπαριθμών 5. Εάν για τον λόγο αυτό το Λαϊκό Κόμμα θα ήθελε να ψηφιστεί ξεχωριστά η τροπολογία 5, τότε εγώ θα ζητήσω παρακαλώ να γίνει χωριστή ψηφοφορία και για την 8. Όμως όλε τι άλλες, εκτός από 5 και 8, μπορούμε να τι ψηφίσουμε αν θέλετε όλες μαζί. Να το το 8 λοιπόν λέει ο Πρόεδρος που ξανά ήρθε στη συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποφέρει κάποιες αποσαφηνίσεις, να μας πει δύο λόγια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία απάντηση μπορώ να δώσω στις ερωτήσεις που αφορούν αυτά τα 15 εκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στη νέα γραμμή του προϋπολογισμού ε, υπό το 2 με τίτλο με επικεφαλίδα ε, κλιματική αλλαγή. Πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα δαπάνηση των χρημάτων αυτών υπό το 2 και επομένως δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα 15 εκατομμύρια ευρώ εκεί που βρίσκονται. Η ιδέα της μεταφοράς των 15 εκατομμυρίων στο 1α για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να καλυφθούν κάποιες ε, προϋποθέσεις. Δηλαδή, εάν ε, υπάρχει ένα όριο τουλάχιστον 13 εκατομμύριων, εκατομμύριων ευρώ στο 1α, έτσι ώστε να μπορέσουν ε, να χρησιμοποιηθούν οι δαπάνες αυτές σε μεταφορά από το 2 και να αυξηθούν οι γραμμές για, την, για το σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης ανάκαμψης. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο περιθώριο στο, στο ε, όριο των, του 1α, τότε θα πρέπει ε, να περιμένουμε πρώτα να γίνει αναθεώρηση των ορίων και μετά των οροφών, των πλαφών και μετά ε, να μπορέσουμε να δούμε εάν μπορούμε να έχουμε αυτή την τεχνική προσαρμογή ε, γιατί ξέρετε ότι έτσι κι αλλιώς ε, βάσει της φύσεως των δαπανών ορίζονται ε, τα διάφορα, οι διάφοροι τομείς και τα διάφορα κεφάλαια και ορίζονται και οι πολιτικές ακριβώς βάσει των δραστηριοτήτων. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν αυτά που ακούσαμε, τις εξηγήσεις που ακούσαμε, κύριε Λαβία, προτείνεται ψηφοφορία κατά τμήματα. Όντως το επιβεβαιώνω. Φαντάζομαι ότι και ο κύριος Γκάιερ ζητάει ψηφοφορία κατά τμήματα ε, για το 8. Προτείνω λοιπόν να ψηφίσουμε on block όλες τις τροπολογίες εκτός από, τις 5, εκτός από την 5 και την 8. Tous les amendements, sauf le 5 et 8. Ε, ψηφοφορία λοιπόν on block εκτός από το 5 και το 8 υπέρ, κατά, τρεις ψήφοι κατά, αποχές, καμία αποχή. Επομένως όλες οι τροπολογίες εγκρίνονται on block. Τώρα τροπολογία 5 του εισηγητού υπέρ κατά. Ένα τμήμα του ΕΛΚ, ε, οι φιλελεύθεροι και κάποιοι άλλοι είναι κατά. Αποχές. Ε, πάντως υπάρχει η πλειοψηφία που εγκρίνει την τροπολογία 5. Τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης, ε, ε, σαφής ε, η υπερψήφιση της τροπολογίας 8. Επομένως, όλες οι τροπολογίες εγκρίνονται, άλλες εγκρίθηκαν, άλλες με πλειοψηφία και άλλες ομόφωνα. Τώρα, τελική ψηφοφορία υπέρ και εδώ πρέπει να καταμετρήσουμε ψήφους. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Επομένως, όλοι οι παρόντες πλην δύο ε, ψήφισαν υπέρ, πλην ε, τριών, συγγνώμη, ψήφισαν ε, υπέρ και δεν υπάρχει καμία αποχή. Τελική άλλη, τροπο... άλλη έκθεση. πρώτη τελευταία ψηφοφορία μάλλον είναι η έκθεση του κυρίου Αλφόνση για τις νήσους του Σολομόντος. Δεν έχουμε ε, καμία τροπολογία, ο εισηγητής είναι υπέρ. Ε, ποιος είναι υπέρ των νήσων του Σολομόντος, λέει ο πρόεδρος. Επομένως, όσοι υπερψηφίσουν, αμέσως θα φύγουν για τα για νησιά του Σολομόντος. Υπέρ, κατά. Δύο ψήφοι κατά παρόλα αυτά. Αποχές. Και εδώ θα πούμε ότι όλοι οι παρόντες πλην δύο εψήφισαν υπέρ. Έκθεση της κυρίας Γιούτα Χάουγκ. Έχουμε εδώ ένα κατάλογο ψηφοφορίας. Από ό,τι μου λένε, οι τροπολογίες Βέρτμαν έχουν αποσυρθεί. 33, 36 και 38. Ο Κέρον θέλει να πάρει το λόγο. θα παίξω το ρόλο της κυρίας Χάουκ σήμερα. Μου ζήτησε να την αντικαταστήσω γιατί κολλείεται. Μου ζήτησε να πω λίγα λόγια ως εξή. Το συζητήσαμε. Αυτό πρόκειται για την συγχώνευση των μεγάλων συστημάτων Schengen, Eurodac και Vis. Υπήρξαν ορισμένε τροπολογίε. Η εισηγήτρια προτείνει μια συμβιβαστική τροπολογία η οποία λαμβάνει υπόψη την υπαριθμό 34, Άλβαρο 35, Κολίνο και την δική της 14 για θέματα καταλήματος προσωπικού κλπ. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, προτείνει προφορική τροπολογία που νομίζω την έχετε μπροστά σας γραπτός, που λαμβάνει υπόψη τροπολογία 26 Βέρτμαν, αλλά και την δική της τροπολογία 15. Επίσης, ήρθε σε επαφή με την Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών, ενημέρωσε ορισμένους συναδέλφους ότι σύμφωνα με την ε, ε, διέρεση αρμοδιοτήτων μεταξύ τη δική μα Επιτροπή και τη Επιτροπή ΛΥΜΕ πρέπει να επαναξεταστούν ορισμένε τροπολογίε. Οι περισσότερε όμω από αυτέ ούτω ή άλλω έχουν αποσυρθεί από την κυρία Βέρτμαν. 33, 36 και 38 έχουν αποσυρθεί από ό,τι βλέπω. Η εισηγήτρια προτείνει η αρχική γνωμοδότηση να ψηφιστεί ολόκληρη μαζί 1 έως 24 τροπολογίες, με εξαίρεση την αμφισβητούμενη 4, ε, η οποία όμως θα καλύπτεται εάν εγκριθεί 28. Κατά τα λοιπά προτείνω να ακολουθήσετε την λίστα ψηφοφορίας. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Σας προτείνω επιμένω, επομένως, αφού δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο, να ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το μπλοκ 1. Τροπολογίες 1 έως 24 εκτός, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως και αναφέρετε και στην ε, λίστα σας, εκτός από τις αμφισβητούμενες 4, 14, 15, υπέρ, κατά, μία ψήφος κατά, αποχές και μία αποχή. Επομένως το μπλοκ 1 εγκρίνεται. Καλύπτεται η τροπολογία 3, αλλά δεν καλύπτεται η τροπολογία 28 του κυρίου Άλβαρο. Ο εισηγητής είναι υπέρ, ψήφι υπέρ κατά αποχές. Η τροπολογία 28 εγκρίνεται, η τροπολογία 4 καλύπτεται από την τροπολογία 28, η τροπολογία 29 καταπίπτει, οι τροπολογίες 5 και 6 καλύπτονται από τον μπλοκ, η τροπολογία 30 Άλβαρο δεν καλύπτεται και η εισηγήτρια είναι κατά, υπέρ της 30 φίλη φιλελεύθερη και ο κύριος Μπόκραους. Ε, κατά. Σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι. Αποχές. Δεν υπάρχει καμία αποχή. Επομένως απορρίπτεται η τροπολογία 30 του κυρίου Άλβαρο. Η 7 καλύπτεται, η 8 καλύπτεται. Τροπολογία 31 Άλβαρο, αλλά με θετική γνώμη του εισηγητού υπέρ, κατά, αποχές. Μία αποχή εγκρίνεται η 31. 32 Βέρτμαν. Πρόκειται για μια τροπολογία η οποία δεν αποσύρεται, είναι συμβατή. Ο εισηγητής δεν είναι υπέρ, ψήφι υπέρ. James Ellis και κάποιοι άλλοι. Κατά. Οι περισσότεροι από ό,τι φαίνεται απορρί... απορρίπτεται τροπολογία. Επόμενη τροπολογία, συμβιβασμός α κεφαλαίο της κυρίας Χάουγκ υπέρ. Κατά αποχές ο συμβασμός α κεφαλαίο εγκρίνεται. Άρα, τροπολογία 15, προφορική τροπολογία της εισηγήτριας, είναι προφορική μεν, αλλά έχετε γραπτό κείμενο μπροστά σας κυρίως η Τσάλ in particular, θα ασχοληθεί με την δυνατότητα κάλυψης των δραστηριοτήτων, ε, κυρίως δε σε περίπτωση που αυτές γίνουν περιτές. Δηλαδή, ε, στην ουσία λέει <laughs> ότι, ε, και είναι μια θαυμάσια απόφαση, ότι εάν κριθεί περιττό, τότε θα καταργηθεί. Άψογα. Προσθήκη λοιπόν αυτής της προφορικής ρυπολογίας υπέρ, κατά, Δύσκολο είναι να είναι κανείς κατά μια τέτοια τροπολογία, λέει ο πρόεδρο. Αποχέ. Συμφωνούμε όλοι λοιπόν ότι όταν κάτι γίνει περιττό θα πρέπει να καταργείται. Τροπολογία λοιπόν 37 Χολμάιερ που δεν καλύπτεται. η εισηγήτρια είναι υπέρ. Υπέρ κατά μία ψήφος κατά. Αποχές καμία αποχή επομένως εγκρίνεται η 38 έχει αποσυρθεί, 20 οι άλλες καλύπτονται. Επανερχόμεθα στην τροπολογία 25 της κυρίας Χολμάγερ πάλι. Η συγκεκριά είναι υπέρ, ψήφι υπέρ, κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 25. Οι άλλες ε, καλύπτονται, εκτός από την τροπολογία 27 του κυρίου Άλβαρο, θετική εισήγηση του, γνώμη του εισηγητού, υπέρ, κατά, αποχές μία αποχή, αλλά η 27 εγκρίνεται. Ε, το ένα καλύπτεται από το μπλοκ 1. Τελική ψηφοφορία υπέρ. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά αποχές. Καμία αποχή. Επομένως όλοι οι παρόντες και ψηφίζοντες είναι υπέρ, πλην τριών που απέχουν. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χάουγκ και βεβαίως τον συνάδελφο που την εκπροσώπησε. Oui, alors, pardon, on n'a pas, pas fini les votes. Δεν τελειώσαμε ακόμα τις ψηφοφορίες, διότι πρέπει να μελετήσουμε ακόμα το πρόβλημα του διορθωτικού προϋπολογισμού 2. Και θα δώσω το λόγο στον ε, εισηγητή μας για το διορθωτικό προϋπολογισμό 2. Και μετά θα του δώσω το λόγο για το πρόβλημα ε, των διορθωτικών προϋπολογισμών 5 ε, και 7. Colleagues, if you remember... Ευχαριστώ πολύ. Ίσως θυμάστε ε, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία και θα θυμάστε φαντάζομαι ότι το κείμενο του Διορθωτικού Προϋπολογισμού 2 περιείχε διάφορα πράγματα τα οποία όμως αφορούσαν τον συνάδελφο Βλαντιμίρ Μάνκα ε, και μέρη ε, και τα θέματα της Επιτροπής που είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Αναγνωρίζοντας βεβαίως ότι το Συμβούλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο να υποβάλει τις προτάσεις εκείνες οι οποίες αφορούν ε, τους άλλους τομείς αλλά και ότι ταυτόχρονα υπάρχει ανάγκη να δοθεί πράσινο φως ε, στις ε, αλλαγές οι οποίες αφορούν την Επιτροπή αποφασίστηκε να διευρυνθεί ε, η αρχική μορφή του 2 και επομένως έχουμε τροποποιητικό προϋπολογισμό που θα δίνει απλώς την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα στον κατάλληλο ε, στην κατάλληλη θέση. Ενώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα και εξ αυτού ε, θεωρώ ότι η Επιτροπή μας μπορεί να υπερψηφίσει την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συμπληρώσω τα λεγόμενα του εισηγητού μας λέγοντας ότι είναι ένα θέμα το οποίο στα πλαίσια του ημερού διαλόγου το είχαμε ήδη εξετάσει. Θεωρήσαμε ε, τότε ότι το Συμβούλιο δεν είχε την πολιτική δυνατότητα να ψηφίσει τον διορθωτικό προϋπολογισμό τον οποίο χρειάζονται ε, και η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών. Όμως, το Συμβούλιο μαζί με την Επιτροπή και ε, απριορεί και υπό την αίρεση της τελικής έκβασης ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου να δεχτεί, λαμβάνοντας υπόψη την ε, ε, μεγάλη ανάγκη, να δοθεί να δοθεί στο ΠΕΡΕΚ, όχι Μπέρες, Body of Current Communications, τέλος πάντων να δώσει σε αυτήν την νέα υπηρεσία, την ΠΕΡΕΚ, ε, την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν θετική ε, ε, γνώμη των τριών οργάνων να δοθούν τα οικονομικά μέσα βάσει του διορθωτικού προϋπολογισμού 2 τα απαραίτητα μέσα ακριβώς όπως πρότεινε και ο εισηγητής μας. Θα ήθελα να κάνω μια προφορική τροπολογία απλώς για λόγους ε, νομικής αποσαφήνισης. Ε, μεταξύ ε, στα, στα, στις παύλες θα πρέπει να βάλουμε και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μεταβατικά μέσα, γιατί, μέτρα, γιατί στον διορθωτικό προϋπολογισμό του 2010 εμείς αναφερόμαστε στην προσωρινή διαδικασία επί της οποίας συμφωνήσαμε τον Νοέμβριο του 2009 στα πλαίσια μια διαθεσμικής συμφωνίας για ολόκληρη τη χρονιά του 2010 αναμένοντας βεβαίως τον την κανονική ε, δημοσιονομική διαδικασία για τα επόμενα χρόνια και επομένως τότε θα πρέπει να γίνει και κάποια προσαρμογή των ημερομηνιών που αναφέρονται στο έγγραφο γιατί ε, μερικές φορές δεν είναι οι σωστές, δεν συμπίπτουν. Πολύ ωραία. επομένω, ε, εάν δεν ζητά κάποιος άλλο το λόγο, να ψηφίσουμε από αυτού του διορθωτικού προπολογισμού 2 υπέρ, κατά, μία ψήφος κατά, αποχές, μία αποχή επίσης. Επομένως ε, εγκρίνεται και συγχαίρω τον εισηγητή. Μια και βρισκόμαστε λοιπόν στους διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Je vais, je vais demander à notre rapporteur θα ζητήσω από τον εισηγητή μας να μας παρουσιάσει την προβληματική, η οποία φαίνεται είναι ε, κοινή για τους διορθωτικούς προεκλογμούς 5 και 7. Χθες το βράδυ είχαμε μια μακρά συζήτηση και με τους συντονιστές για το θέμα αυτό και οι συντονιστές συμφώνησαν ε, με την πρόταση η οποία θα κάνει εξ ονόματός μας τώρα ο εισηγητής. Uh, Σας ευχαριστώ για τον τροποποιητικό προϋπολογισμό 5 δεν αποτελεί πρόβλημα στην αρχική του μορφή και μπορεί να υποστηριχθεί το δυνατόν συντομότερο γιατί καλύπτει τις ανάγκες της Όλαφ. Εμείς είμαστε πάντως διατεθειμένοι να τον υποστηρίξουμε. Δεν ξέρω αν νομικά είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε ή όχι. Να είναι γνωστή δηλαδή η θέση του Συμβουλίου ή όχι. Πάντως ανεξάρτητα από αυτό η θέση μας είναι σαφής ότι δηλαδή τον υποστηρίζουμε. Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, όχι μόνο μεταξύ των συντονιστών, αλλά αν θυμούμε καλά και σε άλλες ευκαιρίες, δηλαδή ότι Θέλουμε οπωσδήποτε να δώσουμε θετικά μηνύματα και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή για να κάνουν κάτι για να ενισχύσουν τη θέση του ευρώ και να είδος εγγύησεως για να υποστηρίξουν εγγυήσεών μάλλον τις χώρες εκείνες οι οποίες βρίσκονται σε άσχημη οικονομική κατάσταση μέσα στην Ευρωζώνη και έξω από αυτήν. Για το λόγο αυτό 60 δισεκατομμύρια, το ποσό 60 δις αναμένεται να λειτουργήσει ως ένα είδος εγγυήσεως για τα δάνεια. Θα θέλαμε πάντως το μήνυμα που θα δώσουμε να είναι θετικό ότι δηλαδή η φιλοδοξία μας να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση είναι κάτι που υποστηρίζουμε. Τώρα πώ να κάνουμε αυτά το δυνατόν συντομότερο. Στη διάρκεια του τριμερού διαλόγου ο πρόεδρο μα έθεσε το θέμα και είπε ότι στον επόμενο τροποποιητικό προπολογισμό μπορούμε να τροποποιήσουμε τον τροποποιητικό προπολογισμό και να κάνουμε και τη δουλειά μα Αυτό δεν είναι πολύ περιπλοκό. Χρειάζεται να προσθεθεί μια νέα γραμμή στον προπολογισμό χωρί χρήματα, κονδύλιο χωρίς να προβλέπετε, να προβλέπετε χρήματα, δηλαδή ένα προσυπόμνηση για τις ε, υποχρεώσεις και ένα PM για τις ε, ε, δαπάνες πλειομών για τις πιστώσεις πλειομών Βέβαια εδώ εκφράστηκαν και κάποιες, κάποιες αντίθετες νομές δηλαδή κυρίως από την νομική υπηρεσία της Κομισιόν, η οποία είπε ότι είναι αντίθετη, διότι είπε ότι μπαίνουμε στα δικά τους δικαιώματα, δηλαδή αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία που είναι όμως προνόμιο της Κομισιόν το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Εμείς απορρίπτουμε την ιδέα αυτή, θεωρητικά, διότι αν είναι έτσι δεν υπάρχει χώρος πλέον να καταθέσει καμία τροπολογία το Κοινοβούλιο. Κάθε ε, ε, τροπολογία αποτελεί ανάληψη μιας πρωτοβουλίας. Νομικά λοιπόν δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Αυτό όμως που συνέβη ή που ίσως στη βάση των ιδεών μας ή των σχεδίων μας είναι ότι η Κομισιόν αντέδρασε γρήγορα και υπέβαλε νέο ε, τροποποιητικό προϋπολογισμό, τον υπαριθμων 7, που είναι ακριβώς αυτό που λέμε, που συζητούμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό σε αυτό το ευαίσθητο θέμα να δούμε πώς μπορούμε να υπερασπιστούμε το ευρώ ως νόμισμα σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς και θα ήταν λάθος να αρχίσει μια δια, διοργανική διαμάχη όπου εμείς και καλά υποστηρίζουμε τη δική μας λύση και απορρίπτουμε την δική τους λύση. Ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν πολύ λάθος. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το χρονοδιάγραμμα, το χρονισμό ας πούμε, το timing, είναι αδύνατον να ψηφίσουμε τώρα τον προπολογισμό υπαριθμών 7, γιατί δεν γνωρίζουμε επισήμω την θέση του Συμβουλίου. Και εγώ ίδιος σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπόρεσα να υποβάλω έκθεση που να υποστηρίζεται από την ομάδα. Όπως είπα όμως μας ενδιαφέρει να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα και στην συνάντηση των συντονιστών υποστηρίχθηκε η ιδέα να γίνει τώρα μια πολιτική ψηφοφορία που θα είναι η έκφραση της ιδέας ότι η παρούσα Επιτροπή Προϋπολογισμών υποστηρίζει την ιδέα να δημιουργηθεί ένα νέο κονδύλιο χωρίς ε, πρικοδότηση, χωρίς να έχει δηλαδή χρήματα, με ένα προσυπόμνηση, προσυπόμνηση για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και για τις πιστώσεις πληρωμών, που θα δίνει όμως τη δυνατότητα όταν θα έρθει η ώρα να μπορέσει να κινητοποιηθεί το σύστημα στο μέλλον. Ελπίζω ότι η επίσημη απόφαση μπορεί να ληφθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Προεπολισμών τον Σεπτέμβρη και μετά να υποβάλουμε τον ε, τροποποιητικό προεπολισμό στην Ολομέλεια. Επ' αυτού χρειάζομαι την γνώμη της γραμματείας, αν μπορούμε να ψηφίσουμε τον amending budget 7 σήμερα ή αν πρέπει να περιμένουμε την θέση του Συμβουλίου. Από τη δική μου σκοπιά δεν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να ψηφίσουμε αν θέλουμε. Και θα σας παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε, στη συνέχεια της αρχικής σας προτάσεως, να προχωρήσετε σε αυτή την πολιτική ψηφοφορία για το θέμα του τροποποιητικού προϋπολογισμού υπαριθμών 7. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Καταλάβατε αγαπητοί συνάδελφοι ότι τώρα δεν σας προτείνω αυτή τη στιγμή νομικής φύσεως τροπολογία όμως να κάνουμε ε, αυτήν την ψηφοφορία έτσι ώστε να ξέρουμε πώς έχει ε, η κατάσταση και ποια είναι η θέση μας απέναντι στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο ε, όσον αφορά τους προϋπολογισμούς, τους amending budgets 5 και 7 γιατί το Συμβούλιο δεν έχει αποφασίσει ακόμα και πρέπει να πούμε ότι πριν την Ολομέλεια θα πρέπει να έχουμε και μία ένδειξη. Και εάν για τον 5 τα προβλήματα δεν είναι πολλά, για τον 7 ε, πραγματικά είναι πολύ σημαντική η κατάσταση, είναι επίγουσα η κατάσταση, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε τι ε, θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, τι μπορεί να κάνει στα πλαίσια των 60 δις ευρώ. Και μάλιστα να σας πω ότι σήμερα το πρωί μάθαμε ότι οι εταιρείες αξιολόγησης ε, ε, ε, έδωσαν μια ακόμα πιο αρνητική θέση στην Πορτογαλία. Υποβίβασαν την Πορτογαλία. Επομένως, ο, αυτός ο μηχανισμός, ε, ο χρηματοπιστωτικός θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θα θυμάστε φαντάζομαι ότι εμείς στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχαμε θίξει το πρόβλημα και όταν η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αυτόν τον χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, είμαστε εμείς που είπαμε ότι δεν προβλέπεται ε, ε, με νομική διασφάλιση αυτή η εγγύηση στα πλαίσια του, των ευρωπαϊκών συνθήκων και επομένως ακριβώς γι' αυτό το λόγο διηθήκαμε στον τροποποιητικό προϋπολογισμό υπαριθμών 7. Έγιναν διάφορες σκέψεις Δηλαδή είτε ε, να κάνουμε κάποια τροποποίηση στον 5 είτε να ενσωματώσουμε τον 5 στο 7. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό τώρα ε, για μας είναι να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Είμαστε αρκετά αριθμοί ε, αυτή τη στιγμή για να στείλουμε ένα καλό πολιτικό μήνυμα. Αφενός προς ε, τις ε, δύο, ε, τα δύο άλλα θεσμικά όργανα και αφετέρου προς την κοινή γνώμη γενικότερα. Ένα μήνυμα που θα λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μια συγκεκριμένη θέση και ότι εν πάση περιπτώσει είναι έτοιμο να περάσει και στην επίσημη απόφαση την επόμενη Ολομέλεια. Ο Σαλβαδόρ και μετά η Ίγκε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, πολιτική αυτή πρωτοβουλία. Θα ήθελα μόνο λίγες διευκρινήσεις, μια και η δημοσιονομική διαδικασία για τους τροποποιητικούς αυτούς ε, προϋπολογισμούς, για τους διορθωτικούς, ε, προβλέπει αρχική ψηφοφορία στο Συμβούλιο, έναρξη προθεσμίας 45 ημερών, προκειμένου να λάβει θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λάβει μια απόφαση και σήμερα ο λάσλο προτείνει μία γραμμή προς υπόμνηση. Κάτι που προϋποθέτει ότι εμείς σε αυτή την προθεσμία των 45 ημερών, αν χρειαστεί, θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε και πάλι αυτό τον διορθωτικό προϋπολογισμό υπαριθμών 7. Αν χρειαστούν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Η σημερινή ψηφοφορία δηλαδή θα μας δέσει τα χέρια ώστε αν παραστεί ανάγκη να μπορέσουμε να υποβάλουμε κατόπιν τροπολογίες στον διορθωτικό προϋπολογισμό 7 εφόσον το δεχτεί το Συμβούλιο με θετική ψήφο. Πολύ σημαντική αυτή η διευκρίνηση και επικροτεί και ο εισηγητής και εγώ άλλωστε. Ingeborg Gressle. Σχεδόν καλύφθηκα, επισημαίνω μόνο ότι έχουμε ανάγκη και από άλλα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε για να στερεώσουμε τη θέση μας στο θέμα αυτού του πακέτου διάσωσης. Γιατί τα όσα κάνει το Συμβούλιο μέχρι τώρα δεν είναι επαρκή ούτε σωστά. Ράιμερ Μπέργκερ. Υποστηρίζω απολύτως αυτά που προτείνει ο Λάσλο Σούριαν αργότερα που θα έρθουμε στην ενδιάμεση έκθεση για την προσαρμογή στην συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ξαναδούμε την ιδέα αυτή ότι υπάρχει το θέμα δηλαδή της περαιτέρω διαδικασίας αλλά και των μελλοντικών ενδεχομένων γεγονότων που θα μας καλέσουν να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην βάση της εμπειρίας ότι είναι κατανοητό μεν ότι η Κομισιόν επιμένει και στον τριμερή διάλογο στην, ε, στο δικαίωμα πρωτοβουλίας της το οποίο υποτίθεται ότι διακυβεύει το Κοινοβούλιο με το PM που ζητάει, το που ζητάει να μην επιμένει στο δικαίωμά της πρωτοβουλίας μόνο απέναντι στο Κοινοβούλιο, αλλά και απέναντι στο Συμβούλιο. Να επιμείνει και να εμείνει και εκεί και όχι να τρέχει από πίσω από το Συμβούλιο το οποίο τη σοφία του έχει αποφασίσει το Α ή το Β. να επιμένει λοιπόν στην επιλογή των σωστών νομικών βάσεων και όχι των ε, πολιτικά πιο ε, ενδεδειγμένων. Είναι ενδεδειγμένο τώρα να βρούμε πάντως πολιτικά μια λύση, ώστε να έχουμε και τη μελλοντική συνεργασία βασισμένη σε μια ξεκάθαρη και υγιή βάση. Merci, Ευχαριστούμε, Ράιμερ. Έχεις δίκιο που έβαλες τα πράγματα στο νέο πλαίσιο. Ο Γκέραν Φέρμ. Μία σύντομη δήλωση. Κανένα πρόβλημα με μια νέα γραμμή προς υπόμνηση. Πολύ σημαντική, απαραίτητο τμήμα της λύσης, αλλά δεν θα προδικάσουμε έτσι την συζήτηση για το πού θα βρούμε τα χρήματα, πού θα βρούμε τα κονδύλια για να ε, τηρήσουμε αυτή την εγγύηση. Πάντως, ε, να θεσπίσουμε μια νέα δημοσιονομική γραμμή προς υπόμνηση δεν μας βρίσκει ενάντια σου. Ωραία. Εύστοχες αυτές οι παρατηρήσεις και σας προτείνω κι εγώ, όπως είπε και ο συγγετής, να ε, κάνω μια πολιτική ψηφοφορία για το σύνολο του τροποποιητικού, των τροποποιητικών προπολογισμών 5 και 7. Ποιος είναι υπέρ δύο ψηφικάτα, αποχές, χωρίς αποχές. Σας ευχαριστώ. Σημαντική πλειοψηφία υπέρ των δύο διορθωτικών προϋπολογισμών 5 και 7, χωρίς νομική αξία βέβαια αυτή η ψηφοφορία και με τις διευκρινήσεις που μας έκαναν οι συγητές και οι προλαλήσαντες, και οι προλαλήσαντες. Μάλιστα αργότερα θα έχω γεύμα εργασίας με την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και θα έχω την ευκαιρία να επισημάνω πολλά και διάφορα στην Κορεπέρ και για την δημοσιονομική διαδικασία του 2011, όπως είπαμε χθε, και για τη θέσπιση αυτού του μηχανισμού, αλλά και τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ναι και βλέπω σε φόρμα τον εισηγητή και έχει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη της Επιτροπής προπολογισμού πώς θα μπορούσε να μας παρουσιάσει και τις μεταφορές πιστώσεων. Για να δούμε εντάχει τι μεταφορέ. Από ό,τι βλέπω έχουμε πέντε προτάσεις μεταφοράς. Καταρχήν, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τη 19, την 23 και την 25. Δεν είναι καθόλου επίμαχες και τις στηρίζω. Το ίδιο ισχύει σχεδόν και για την 27. αλλά δυσαρεστούμαστε κάπως γιατί δεν είναι καλές οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πιστώσεις πληρωμών. Γιατί πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει τη δική μας προθυμία ή ετοιμότητα να στηρίξουμε τις αιτήσει μεταφοράς πιστώσεων αλλά νομίζω ότι και εκείνη μπορεί να βελτιώσει λίγο τον τρόπο εργασία τη. Συνήθω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει εντάξει, θα τις δεχτούμε την τελευταία στιγμή και σίγουρα το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Είναι κάτι συνηθισμένο. Πάντως, δεν έχω αντίρρηση να υποστηρίξουμε αυτές τις μεταφορές πιστώσεων, Και η τελευταία αίτηση που είναι το 35, αυτό είναι όντως κατεπήγον. Ανέκυψε πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, αφορά 40 εκατομμύρια για την ενίσχυση της Γιούνρα στην Παλαιστίνη και την Παλαιστίνη. Είναι πραγματικά κατεπήγον αυτό το αίτημα Γι' αυτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε δεόντως και με ελαστικότητα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Προτείνω να ψηφίσουμε από κοινού και τις πέντε της μεταφοράς πιστώσεων θετικά. Ευχαριστώ. Φυσικά δεν έχουν αντίρρηση οι ομάδες. Ε. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Υπήρξαν κάποιες ανακρίβειες στο Κόμπου νιούς. Εσείς μας δώσετε πάντως ε, τους ακριβείς κωδικούς των μεταφορών. 19, 23, 25 και 27. Τις έχετε στο φάκελο, συν την 35 της συμμεταφοράς πιστώσεων, που όπως μας είπε ο εισηγητής είναι η πιο πρόσφατη και αφορά ένα συμπλήρωμα ενίσχυσης προς την Παλαιστινιακή Αρχή και τη Γιούνρα. που δίνει συνέχεια στη χθεσινή μας ακρόαση με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής Σαλάμ Φαγιάτ. Συμφωνούμε με τους αριθμούς της μεταφοράς πιστώσεων, έτσι. Να ψηφίσουμε από κοινού προτείνει εισηγητής. Μήπως υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ποιος είναι υπέρ των πέντε μεταφορών πιστώσεων. Κατά. Αποχές. Τρεις ήταν οι ψήφοι κατά. Δεν υπάρχουν αποχές. Σας ευχαριστώ και συγχαίρω τον εισηγητή μας που για μια ακόμη φορά έτυχε τη ε, υποστήριξη τη Επιτροπής Προπολογισμών. Ίγκε. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε. Άλλη μια μεταφορά. Την ΤΕΚ 16. Την οποία είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά. Για μελέτες. Και υπήρχαν και ορισμένες ερωτήσεις την οποία, τις οποίες απάντησε με επιστολή του προς εσάς ο Γενικός Διευθυντής της Κομισιόν κ. Ζανζάν. Θα θυμάστε την ιστορία με τα έπικα της IKEA. Επίσης 150, 155 εκατομμύρια για μελέτες για την ηλεκτρονική τεχνολογία. Αυτά τα αφαιρεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μειώνονται δηλαδή οι μελέτες κατά 1500 από το 2005 με το 2008. Μα υπάρχει κάποια αξιοπιστία πλέον στα δεδομένα της Κομισιόν. Και εν πάση περιπτώσει τι ερμηνεία να δώσουμε. Δηλαδή τους πιάσαμε και τώρα απλώς τα αποσύρουν. Θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα πράγματα για την αξιοπιστία των δεδομένων τους, εάν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, εάν μας έχουν γράψει οτιδήποτε για τα θέματα αυτά. Και εφόσον ήταν μελέτες, αφού ήταν δηλαδή στη γραμμή του προπολογισμού οι δαπάνε αυτές για ηλεκτρονική τεχνολογία ως μελέτες και τώρα μας λένε ότι ήταν ασφαλμένη η καταχώρηση αυτή. Ε, τέλος πάντων, από πού πληρώθηκαν αυτά. Όταν δηλαδή καταχωρούν στα λογιστικά βιβλία μελέτες οι οποίες μετά αποδεικνύουν ότι δεν ήταν μελέτε, πρόκειται για σοβαρή παραβίαση του δικαίου. Θέλω, εν πάση περιπτώσει, να στείλω ορισμένε ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Ίγκε. Πολύ εύστοχη ερώτηση. Το σημείωσε η Ευρωπαϊκή η Επιτροπή μας μάλλον και φαντάζομαι θα σα ε, απαντήσει η προφορικός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά όμω την συνεδρίασή μα, γιατί ελάχιστος χρόνο μα έχει μείνει και έχουμε πολλά σημεία στην ημερήσια διάταξη. Πάντως αν δεν σα ικανοποιήσουν οι απαντήσει της Ευρωπαϊκής τότε θα συμπεριλάβουμε αυτό το σημείο στην επόμενη μα ε, συνεδρίαση. Ο Λάζλο είναι ικανοποιημένο και μπορεί να ξεκινήσει τι διακοπές του γιατί εργάστηκε πολύ καλά. Επόμενες μεταφορές πιστώσεων θα μας παρουσιάσει ο Βλέντιν Μάνκα. Εδώ έχουμε πολλές μεταφορές, κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ. Έχουμε αρκετές μεταφορές στην τελευταία συνεδρίαση είπαμε όλο το πακέτο του οριζόντιου υποθυνομικού το 45% ε, για την μετάφραση θα το δούμε σήμερα. Θα θυμούνται ίσως οι συνάδελφοι ότι προβλέψαμε ένα οριζόντιο αποθεματικό 5% γιατί το 2006 το ελεκτικό συνέδριο επισήμανε ένα πρόβλημα με τα αποθεματικά της ε, διασυνοριακής συνεργασίας για τη μετάφραση. Και υπάρχει το θέμα της εξωτερικής ανάθεσης ε, της μετάφρασης, χωρίς ε, να εξακριβώσει αν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα έχουν αποθέματα σε, σε θέματα μετάφρασης. Γι' αυτό είπαμε μόνο 5% αποθεματικό και μόνο αν αποδείξουν θεσμικά όργανα ότι χρησιμοποιούν και αξιοποιούν την ε, ε, διαθεσμική συνεργασία θα αυξήσουμε το αποθεματικό και ε, θα τα αφαιρέσουμε από το αποθεματικό. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η οργανική συνεργασία έχει βελτιωθεί από την άποψη αυτή και υπάρχουν αρκετά εργαλεία και μηχανισμοί για την βελτίωση, αναβάθμιση των μεταφράσεων. Έχουμε το σύστημα σε μια τεράστια βάση δεδομένων με εκφράσεις ε, και ολόκληρες προτάσεις μερικές φορές που χρησιμοποιούνται σε έγγραφα που είναι προς μετάφραση. Οπότε προτείνω κατάργηση του αποθεματικού, αλλά διαπίστωσα ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα. Ίσως, ίσως θα θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι ότι πολύ συχνά στην ημερήσια διάταξή μας έχουμε μεταφορές που μεταφράζονται μόνο σε δύο γλώσσες, ε, στα γαλλικά και τα αγγλικά. Και αν εγκριθούν ε, έγγραφα σε μία από τις δύο γλώσσες, μετά μεταφράζονται στις υπόλοιπες. Αλλά μένουν να χρησιμοποιεί τα, τα έγγραφα αυτά. Ενώ άλλες φορές χρειαζόμαστε στην ημερήσια διάταξη έγγραφα μεταφρασμένα και δεν τα έχουμε γιατί εξαντλήσαμε το δυναμικό μας σε μετάφραση περιττών ουσιαστικά εγγράφων. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ίσως να το φροντίσουμε στον επόμενο προπολογισμό του 2011. Γιατί δεν είναι αποδοτικός αυτός και αποτελεσματικός τρόπος εργασίας, ούτε γίνεται ορθολογική χρήση των μεταφραστικών μας δυνατοτήτων, μια και μεταφράζουμε περί τα έγγραφα και δεν μας μένει δυνατότητα για μετάφραση των χρήσιμων. Ή, το χρησιμοποιείται αυτό με δυναμικό αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ΟΚΕ, την Επιτροπή Περιφερειών και αν συμφωνεί και ο Λάσλο για το τμήμα της Επιτροπής μπορούμε να άρουμε το αποθεματικό, να το απελευθερώσουμε. Πάντως το ζητούμενο είναι η αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των μεταφράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και περιμένω το σχόλιο των συναδέλφων. Ε, ε, Λάσλο, και Σούριαν, συμφωνείτε με την πρόταση του Βλάντιμιρ Μάνκα για απελευθέρωση του αποθεματικού του 5% που ίσχυε οριζόντια για το Κοινοβούλιο, την Επιτροπή την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών. και αντιστοιχεί στο μεταφορά πιστώσεων 23 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπέρ. Ωραία, μπορούμε να ψηφίσουμε. Για την κατάρριση του αποθεματικού Υπέρ, κατά. Αποχές, μία ψήφος κατά. Ωραία. Ο κύβος ερήφθη. Ο κύριος Μάνκα έχει τρία ακόμη αιτήματα μεταφοράς πιστώσεων, έξι και επτά για το Κοινοβούλιο και τρία για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω με την μεταφορά τρία για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. οι αριθμοί των ε, τραπεζικών μεταφορών έχουν ε, μειωθεί. Ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κέρδισε κατά κάποιο τρόπο 11 εκατομμύρια, αλλά χρειάζεται τα χρήματα αυτά και πρέπει να πω ότι πρέπει να γίνουν κάποιες μελέτες για τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά. Ε, υπάρχουν επίσης εκκρεμίε υποθέσεις και επομένως αυτά ε, τα... Ε, αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως, ο εισηγητής δεν προτείνει ε, να ε, χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά, να δοθούν τα χρήματα αυτά έτσι ώστε συστηματικά να αποφαίνεται θετικά υπέρ του Κοινοβουλίου. Ούτε το υπονοεί. Ωραία. Να ψηφίσουμε λοιπόν για την μεταφορά αυτή υπέρ, κατά, αποχές, δύο αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Δύο τελευταίες μεταφορές πιστώσεων. έξι και επτά, αφορούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επομένως μπορούν να παρουσιαστούν και να ψηφιστούν από κοινού. Κύριε Ισηγητά, ευχαριστώ. Ναι, όντως μπορούμε να ψηφίσουμε για αυτές τις δύο μεταφορές μαζί. Ε, πρόκειται για θέματα τεχνολογίας της ε, πληροφορίας ε, και είχε συζητηθεί το θέμα αυτό το προηγούμενο Οκτώβριο και πρέπει να πω ότι εξ του προεδρίου είχα υποβάλει το ποσό των 8 εκατομμυρίων ως αποθεματικό για τις τεχνολογίες πληροφορίας και Ζήτησα να υπάρξει στρατηγική ε, σχετικά με το θέμα αυτό και βεβαίως εάν υπάρξει στρατηγική τότε θα αρθεί ε, το αποθεματικό. Έξι από τα οκτώ εκατομμύρια θα πρέπει να συζητηθούν σήμερα και νομίζω ότι ε, τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις έχουν καλυφθεί και επομένως μπορεί να αρθεί αυτή η επιφύλαξη για τα έξι από τα οκτώ εκατομμύρια. Τώρα, όσον αφορά τα 6,2 εκατομμύρια ευρώ, πρόκειται για χρήματα ε, που αφορούν τους υπαλλήλους, το προσωπικό και νομίζω ότι θα πρέπει να υπερψηφιστούν και οι δύο μεταφορές. Ευχαριστώ. Τώρα, εάν ε, ε, κάποιος ε, από τους συναδέλφους θέλει να υποβάλει κάποια ερωτήματα ή κάποιοι που γνωρίζουν καλύτερα το τομέα της πληροφορικής, αν θέλουν να μας διευκρινίσουν κάτι, βεβαίως μπορούν να το κάνουν. Πρόεδρος, ωραία, δεν βλέπω να ζητά κάποιος το λόγο, επομένως ψηφίζουμε τις δύο μεταφορές μαζί. Υποβάλλω λοιπόν προς ψήφιση τις προτάσεις του εισηγητού Αμπλοκ υπέρ, κατά, ευχαριστώ πολύ, δύο ψήφι κατά, αποχές, καμία αποχή και επομένως αποφασίσαμε θετικά υπέρ των δύο ε, αυτών θεμάτων. Επομένως εξαντλήσαμε τα θέματα ε, των μεταφορών πιστώσεων και προτείνω τώρα να περάσουμε σε μια άλλη ψηφοφορία που μας ζητάει η Μόνικα Χολμάγερ. αφορά το θέμα 25, την κτηριακή πολιτική δηλαδή των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζετε πλέον την διαδικασία του άρθρου 179 παράγραφος 3, βάσει του οποίου μάλλον βάσει της οποίας ε, κάθε φορά που ε, γίνεται πρόταση για κάποιο νέο κτίριο η Επιτροπή μας θα πρέπει να αποφανθεί για το κατά πόσον θα γνωμοδοτήσει. Επομένως, βρισκόμαστε τώρα στην πρώτη φάση. Η κυρία Χολμάγερ θα μας μιλήσει για ένα ε, σχέδιο που αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου ε, Νόσων στην Στοκχόλμη. Εάν θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, θα μας το πει. Ή διαφορετικά θα μας πει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Θα μας πει λοιπόν την άποψή της. Και βεβαίως, εάν θεωρήσει ότι πρέπει να ενδιαφερθούμε για το θέμα αυτό, τότε θα προχωρήσουμε ε, σε συζήτηση επί της ουσίας και εις βάθος ε, της εκθέσεώς της και αυτό θα γίνει βεβαίως σε μια επόμενη συνεδρίαση. Και να πω αμέσως και για τα πρακτικά αλλά και για την ε, ίδια την υπηρεσία. Να πω λοιπόν ότι η διαδικασία του άρθρου 179 παράγραφος 3 μας επιβάλλει πολύ ε, στενά χρονικά περιθώρια, τα οποία δεν μπορούμε να σεβαστούμε μέχρι την επόμενη συνεδρίασή μας. Όμως υπάρχει μια συμφωνία κυρίων βάσει της οποίας ε, θεωρείται ότι η θερινή περίοδος ε, αφαιρείται από την προβλεπόμενη περίοδο. Βέβαια αν υπολογίσουμε ότι οι καλοκαίρινες διακοπές για το κοινοβούλιο είναι τρεις μήνες, επιμικίνεται λίγο. Εν πάση περιπτώσει, Μόνικα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τα διευθυνιστικά εισαγωγικά λόγια. Πρόκειται για ένα κτίριο του οργανισμού ECDC που ασχολείται με πρόληψη ασθενειών, νόσων κλπ. Πρόκειται για έναν από τους οργανισμούς που ιδρύθηκε το 2005 και από το 2005 έχει ενισχυθεί σημαντικά. Σε αυτό αναφέρομαι. Υπάρχουν ένα αριθμό οργανισμών που μεγαλώνουν και μεγαλώνουν και εμείς δεν έχουμε απολύτως κανέναν έλεγχο για το πόσο μεγαλώνουν και με ποιο ρυθμό. Θα αποκτήσει λοιπόν μέχρι το 2011 κατά πεσευθενότητα ο οργανισμός αυτός 400 συνεργάτες και χρειάζεται χώρο Προτίθενται λοιπόν να μισθώσουν στην έδρα τους που βρίσκεται κοντά στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και άλλους χώρους. Επίσης να ανεγείρουν νέο κτίριο που θα ανεγείρει ο εκμισθωτής που είναι η Ακαδέμισκα Χις και που είναι ε, ιδιοκτησία του Σουηδικού Δημοσίου. το νέο κτίριο θα κτιστεί ε, δίπλα στο υφιστάμενο. Το 2005 άρχισαν με την μίσθωση δύο κτίριων. Από το 2008 μισθώθηκε και νέο κτίριο όπου δεν ζητήθηκε γνώμη της αρχής ε, του προϋπολογισμού. Είναι όμως δεσμευτικό. Εάν θελήσουμε να φύγουμε θα μπορούσαν να είχαν επιλέξει και ένα άλλο κτίριο αλλά αυτό δεν είναι πλέον δυνατόν διότι βρισκόμαστε σε μια δέσμευση. Εάν επιλέξουμε τώρα άλλο κτίριο από αυτό που μας προτείνεται, καλούμαστε να πληρώσουμε ποινικέ ρήτρε για μια οκταετία. Δηλαδή θα χρειαστεί να πληρώσουμε όλα τα μισθώματα μέχρι το 2018. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για την αρχή του προπολογισμού, διότι δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε με την πρόταση που μας γίνεται, διότι αν δεν συμφωνήσουμε είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε επί 8 έτη μισθώματα και έτσι χάνουμε την ευκαιρία, για παράδειγμα, να ανιμιστώσουμε ένα άλλο κτίριο υπό ευνοϊκότερου όρου. Πρόκειται για ένα θέμα όπου εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να το καταστήσουμε απόλυτα σαφές σε μια γνωμοδότησή μας τον Σεπτέμβριο, διασυνδέοντάς το και με προβλήματα που έχουμε με άλλους ε, οργανισμούς. Και διευκρινίζοντα ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι απολύτω απαράδεκτη. Δεν μπορούν να μα θέτουν πρώτα τελεσμένων γεγονότων με τρόπο ώστε να μην μπορούμε πλέον να λάβουμε καμία άλλη απόφαση. Σχετικά με το κόστος τώρα για το 2009 το κόστος ανέρχεται σε 1,6 εκατομμύρια. ανά τετραγωνικό μέτρο 197 ε, ευρώ. Όπως είπα, η σύμβαση μισθώσεως φτάνει μέχρι το 2018 και αν δεν καταγγελθεί ένα έτος πριν θα ανανεωθεί για άλλα τρία έτη. Αυξάνει όπως είπε ο αριθμός των συνεργατών, βολεύονται τώρα με κοντέινερ και άλλα τέτοια πράγματα που βέβαια δεν μπορεί να αποτελέσει ικανοποιητική λύση στο δινεκές. Νέα σύμβαση χρονομίσθωσης υποτίθεται ότι θα υπογραφεί για το νέο κτίριο και στη νέα σύμβαση θα, να, θα περιληφθεί υποτίθεται και μια ρήτρα break-up Μέχρι τώρα στις συμβάσεις δεν έχουν περιληφθεί ρήτρες break-up. Το καλό για το κτίριο είναι ότι ολόκληρος οργανισμός η e CDC θα μπει μέσα σε ένα κτίριο το οποίο είναι και καλά δομημένο. Ε, γίνονται προσπάθειες ε, να εξορθολογιστεί η χρήση των χώρων ώστε να μειωθούν τα τετραγωνικά μέτρα. Στο μέλλον δεν θα έχουμε κόστος μονάχα 1,6 εκατομμύρια αλλά 2,9 από το 2014 λοιπόν θα χρειαστούν 1,2 εκατομμύρια παραπάνω. Το μέσο μίστομα θα ανέλθει στα 263 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Και όπως είπα συνολικά θα ανέλθει το, το οργανόγραμμα σε 400 θέσεις. Το 2013 προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι κατασκευές αυτές και η ε, νέα, ε, η νέα μίσθωση θα αρχίσει από το 2014. Μετά εδώ μπαίνει και ένα δεύτερο πρόβλημα. Ο ίδιος ο οργανισμός λέει ότι το μέσο μίσθωμα είναι 1500 σουηδικές κορώνες ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχω βέβαια εδώ τα νούμερα στις Σουηδικές κόρονες μπροστά μου, γι' αυτό σας τα λέω έτσι. Η, το, το μέσο μίστομα είναι 2.350. Βέβαια, αυτά λέει η CDC. Αν δούμε τώρα την γνωμοδότηση της ε, Richard Ellis που είναι μια μεγάλο ένας μεγάλος οργανισμός ε, CB Richard Ellis. με σιτικό γραφείο δηλαδή. Αυτά, αυτά τα νούμερα που μας δίνει δείχνουν ότι είναι πάνω από τον μέσον όρο των μισθωμάτων αυτό που πληρώνει η CDC. Λοιπόν, πρόκειται για πρόβλημα. Η πρότασή μου είναι, για τον λόγο αυτό, αφενός γενικά για τους οργανισμούς και ειδικά για την ECDC να συντάξουμε μια γνωμοδότηση μέχρι τον Σεπτέμβριο που θα διαβιβάσω και στους συνεισηγητές για να καταστήσουμε σαφές και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι πάντοτε σημειώνονται περιπλοκές με τους οργανισμούς είτε δηλαδή δεν τηρούνται ε, τα είτε δεν τηρούνται οι όροι των ε, αναθέσεων ή των διαγωνισμών ή Μα προσφέρει για παράδειγμα τώρα η Σουηδική κυβέρνηση ένα κτίριο το οποίο είναι θαυμάσιο πραγματικά, είναι πάρα πολύ καλά φτιαγμένο ε, και από άποψη περιβαλλοντική, εξοικονόμηση ενέργεια κλπ. Έχουν κάνει τα πάντα πραγματικά. Εκεί δεν μπορεί να πει κανεί ότι θα εγκατασταθεί ο οργανισμό σε ένα άσχημο κτίριο. Μπαίνει σε ένα πολύ καλό κτίριο. Αλλά εν τέλει. Είναι ασυντόνιστη η ανάπτυξη αυτού του οργανισμού και η ε, κατάληψη, εγκατάστασή του μάλλον σε ε, κτίρια. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσετε να συντάξουμε μια γνωμοδότηση για τον Σεπτέμβριο, την οποία όπως είπαμε, κάθε λεπτομέρεια θα ε, υποβάλω στους συνεισηγητές. Σας ευχαριστώ για την πάρα πάρα πολύ ακριβή παρουσίαση του θέματος. Κύριε Γένσεν. Όχι, δεν έχω ερώτηση. Υποστηρίζω την εισηγήτρια. Νομίζω ότι έχει εργαστεί καλά. Νομίζω επίσης ότι έχει διαρθρώσει την εργασία της, έχει συντάξει και ένα ερωτηματολόγιο. Και αυτό είναι καλό, για να γνωρίζουμε, να γνωρίζουν και όλοι δηλαδή, τι θα αντιμετωπίζουν. Η γνωμοδότηση είναι σωστή. Είναι ζήτημα αρχής. Ίσως στην Στοκχόλμη να έγιναν πιο συμπτωματικά τα πράγματα από ό,τι αλλού. Αλλά οι εμπειρίες μου δείχνουν ότι τέτοιες περιπτώσεις ξεπηδούν ξανά και ξανά. Άρα χρειάζεται μια πιο συγκεκριμένη και βασική προσέγγιση, βασισμένη σε κάποιες βασικές αρχές. Που άλλωστε είναι μια προσέγγιση που ακολουθούμε και στην Διαθεσμική Επιτροπή για τους Οργανισμούς Αυτό αφορά και χρήση άλλων κτίριων. Νομίζω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία είναι πολύ ορθή και την υποστηρίζω. Ευχαριστώ κύριε Γένση. Ο κύριος Μπούκρος. Σύντομο σχόλιο. Υποστηρίζω απολύτως και την Μόνικα Χολμάιερ και την Αν για το θέμα. Κάθε φορά που έχουμε μπροστά μας ένα θέμα ακινήτου, βλέπουμε κάποιες ανομαλίες δεν γίνονται τα πράγματα με διαφανή τρόπο καθόλου. Υπάρχουν αρκετές ανομαλίες όπως είπα. Τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δαπανώνται με αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν άπαξ και διαπαντός να εγκρίνουμε την μέθοδο που προτείνει η συγκήτρια να λάβουμε υπόψη ότι μιλούμε για τεράστια ποσά και αν αυτά δεν δαπανώνται με σωστό και σόφρονα τρόπο, θα κληθούμε εν τέλει να είμαστε πολιτικά υπόλογοι γι' αυτά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι όντως η εισηγήτριά μας ε, έχει απόλυτο δίκιο και πέρα από τη συγκεκριμένη περίπτωση αυτής ε, της ε, υπηρεσίας το ζήτημα θα πρέπει να τεθεί γενικότερα και βεβαίως να τεθεί υπόψη του, της Επιτροπής για αυτές τις ε, υπηρεσίες. Τώρα, ε, και όσον αφορά αυτήν την ε, συγκεκριμένη περίπτωση της υπηρεσίας για την καταπολέμηση νόσων και έλεγχο, πρόληψη έλεγχο, ε, είτε θα πρέπει να μας πούνε, ξέρετε δεν κάνει καλή δουλειά, άρα έχουμε όλο και περισσότερες ασθένειες, άρα δεν έχει έννοια να τους δίνουμε χρήματα, είτε κάνουν πολύ καλή δουλειά, άρα πρέπει να τους δώσουμε πιο πολλά χρήματα. Ε, πρέπει να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια ε, ήταν ένας άνθρωπος στα Ηλίσια Παιδεία ε, και έλεγε εγώ έχω τη μαγική, <laughs> έχω τη, μαγική σκόνη η οποία απομακρύνει τους ελέφαντες και το πράγμα τι δεν την κάνουμε αφού δεν έχει ελέφαντες μα είδατε πόσο αποτελεσματικός είμαι και πόσο αποτελεσματική είναι η σκόνη. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι κάπω έτσι βρισκόμαστε εδώ. Εν πάση περιπτώσει, η εισηγήτριά μα προτείνει να γνωμοδοτήσουμε. Άρα ψηφίζουμε επί τη προτάσεω τη εισηγήτρια. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά αποχές. Επομένως η κυρία Χολμάιερ θα γνωμοδοτήσει. Τώρα, έχουμε μία μικρή έκθεση ε, του κυρίου Κάλφιν πριν να ολοκληρώσουμε με, μεγαλειώδη τρόπο με τον κύριο Μπέγκε. Πρόκειται ε, για την νομική βάση για την μπανάνα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για τη νομική βάση της μπανάνας. Είναι επίγον το θέμα, γιατί θα πρέπει να εγκριθεί η γνωμοδότηση αυτή τη 13η Σεπτεμβρίου και επομένως ο Ιβο Κάλφιν θα πρέπει να μας παρουσιάσει την πρότασή του και τον ευχαριστώ κιόλας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για κανονισμό τροποποίησης ε, του κανονισμού ε, και δεν αφορά τις μπανάνε, αφορά τις ε, παραγωγέ χώρες. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να υποβάλω. Πρώτον, ότι υπάρχει ένας πολύ σωστός, ορθός λόγος που οδηγεί σε αυτήν την απόφαση η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, επί σειρά ετών ε, στηρίζει τις εξαγωγές χώρες, δηλαδή τις χώρες ΑΚΕ. Όμως, μεταξύ υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες υπέβαλαν στον ΠΟΕ αυτήν την στήριξη με το σκεπτικό ότι αντιτίθεται στις ορθές πρακτικές εμπορίου, ο ΠΟΕ απεφάνθη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως ε, παραβιάζει την αρχή της ε, ισότητας και επομένως ε, από φέτος δεν μπορεί πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει οποιαδήποτε επιδότηση εξαγωγών σε αυτές τις χώρες παραγωγές μπανάνας. Ε, βεβαίως σιγά σιγά οι χώρες αυτές άλλαξαν ε, και το προφίλ της οικονομίας τους και της βιομηχανίας τους. Ε, αλλά εν πάση περιπτώσει όπως και να έχουν τα πράγματα, προτείνω εμείς να πάρουμε σαφή θέση γιατί λόγω της απόφασης του ΠΟΕ πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο στήριξης των χωρών αυτών. Δεύτερο πρόβλημα έγκυται στην πρόταση του Συμβουλίου και της ε, Κομισιόν για τον τρόπο ε, στήριξης ε, αυτής της δραστηριότητας. Το Συμβούλιο λοιπόν απορρίπτει και πρόκειται για απόφαση για τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι το 2013 ε, μιλάμε για 150 εκατομμύρια και επομένως το Συμβούλιο ε, απορρίπτει οποιαδήποτε χρήση εργαλείου ε, ευελιξίας, μηχανισμού ευελιξίας μάλλον, για την στήριξη των μέτρων αυτών. Και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να έχουμε κάποια, να έχουμε κάποιον συντονισμό χρήσης αποθεματικού με εφαρμογή μέτρων ευελιξίας εμείς θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Δύο επιλογές έχουμε. Εάν ε, ήταν προβλέψιμο δεν θα χρειαζόμαστε κανέναν μηχανισμό ε, ευελιξίας, αλλά τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είχε προβλέψει μέτρα στήριξης της μπανάνας στον κανονικό προϋπολογισμό, γνωρίζοντας την απόφαση του ΠΟΕ. Αυτό όμως δεν συνέβη έτσι κι αλλιώς. Επομένως, η Επιτροπή προτείνει την συνέχιση της ε, χρηματοδότησης πέρα από τις ε, ε, συνήθεις πρακτικές του προϋπολογισμού, εκτός προϋπολογισμού, εν πάση περιπτώσει. Σε αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθούν, θα χρησιμοποιηθούν οι μηχανισμοί ευελιξίας και αυτό θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε γιατί θα θεωρηθεί ότι το μέτρο είναι έκτακτο και απρόβλεπτο. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη υπάρχει αντίφαση μεταξύ της πρότασης του Συμβουλίου και της Κομισιόν και το Συμβούλιο δηλαδή δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί η ευελιξία, θα πρέπει να κάνουμε δικιά μας πρόταση. Προτείνω να ε, ε, γυρίσουμε στην Επιτροπή όλη την πρόταση και να ζητήσουμε να ε, προτείνει διαφορετικό καταμερισμό των πηγών χρηματοδότησης. Δηλαδή, Εάν κάτι συμβαίνει, ε, αν συμβεί κάτι απρόβλεπτο, τότε να καλυφθεί από τον μηχανισμό ε, ευελιξίας και ε, να μην χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή χρήση του αποθεματικού ή των περιθωρίων. Ξέρω ότι ενδεχομένως το Συμβούλιο δεν θα δεχτεί πάρα πολύ εύκολα την πρόταση, αλλά τουλάχιστον η απόφαση αυτή θα ευθυγραμμίζεται με όλες τις αποφάσεις που έχει λάβει το Κοινοβούλιο και βεβαίως και πρόκειται για μια προσέγγιση αρχής ε, η οποία είναι ορθότερη. Και εάν ε, έχουμε κάποια περίπτωση ε, απρόβλεπτων γεγονότων τότε να προστρέξουμε στον μηχανισμό ευελιξίας. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να, να γίνει κάποια διαπραγμάτευση μεταξύ Κομισιών και ε, Συμβουλίου και οπωσδήποτε να δοθεί ε, καταμερισμός των ε, χρηματοδοτήσεων και των πόρων χρηματοδότησης. Εν πάση περιπτώσει, επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 50% τουλάχιστον των χρημάτων που προβλέπονται για την στήριξη των παραγωγών μπανάνα στο χώρο και προβλέπεται να δοθεί φέτος και επομένως ε, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση. Βεβαίως ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και γενικότερα το πρόβλημα της χρηματοδότησης αυτών των, ε, χωρών και αυτών των παραγωγών. Εν πάση περιπτώσει έχουμε συζητήσει και με τους άλλους συναδέλφους οι οποίοι συμφωνούν και με, τις, με την πρόταση αυτή η οποία ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες αποφάσεις του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι εάν υπάρξουν απρόβλεπτα γεγονότα, τότε να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμό ευελιξία. Διαφορετικά, εάν δεν προβλέπονται τέτοια απρόβλεπτα γεγονότα, να είχαν προβλέψει, να μην είχαν προβλέψει τον μηχανισμό ευελιξία. Ευχαριστώ. Όντω, συζητήσαμε για την μπανάνα Κοιτάξτε, απλώ ξεφλουδίζουμε την μπανάνα διαφορετικά, λέει ο πρόεδρο. Πότε από τη μία, πότε από την άλλη πλευρά. Έχουμε μία διελκυστίνδα εδώ και το είπαμε και στο τριμερή διάλογο ε, μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή βρίσκεται κάπου στη μέση. Αρχικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε πλήρη χρηματοδότηση με το μέσο ελαστικότητας όπως μας είπε ο εισηγητής. Το Συμβούλιο ήθελε 100% από τη μεταφορά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια ενδιάμεση πρόταση, μια χρυσή τομή, που όμως δεν ήταν αρκετά ακριβωδίκη κατά τη γνώμη μας. Υπάρχει λοιπόν μια διελκυστίδα. Αλλά όπως είπε και ο συγκητής μας, έχουμε συμφέρον για μια γρήγορη λύση. Δεν θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο βάρος των χωρών αυτών που εις βάρος των χωρών που δικαιούνται αυτή την ενίσχυση. Εμείς είμαστε υπέρ και της ιδέας της ενίσχυσης, της αρχής, ε, του ποσού και θέλουμε ένα χρονοδιάγραμμα καταρτισμένο το συντομότερο δυνατό. Η πρόταση αυτή δεν είναι ούτε για να κερδίσουμε ούτε για να χάσουμε χρόνο, αλλά για να καταλήξουμε σε έναν τρόπο χρηματοδότησης που κατά τη γνώμη μας είναι ο πιο σωστός. Η Αν Γένσεν ζήτησε το λόγο. Συμφωνώ, συμφωνώ ότι δεν παίζουμε με το χρόνο εδώ. Γιατί ίσα ίσα η Επιτροπή Ανάπτυξη σας κυπήσει να επιληθεί το πρόβλημα τη μπανάνα το συντομότερο δυνατό. Χρειάζεται το εργαλείο, λένε, στην ανάπτυξη. Δεν είμαστε κατά του εργαλείου και του μηχανισμού. Αλλά συμφωνώ με τον κύριο Κάλφιν ότι αυτός είναι ο ορθός τρόπος δράσης και πραγματικά είναι αποτροπιστικό αυτό. Έπρεπε είτε να το συμπεριλάβουν στο προπολογισμό και θα ήταν έκπληξη ή να χρησιμοποιηθεί το μέσο ελαστικότητας. Αυτές είναι οι δύο ακραίες θέσεις. Βέβαια η Επιτροπή πάντα βρίσκει μεταφορές από προπαρασκευαστικές δράσεις όπως το πρόγραμμα για τον αύξηνο πόντο για επίσης μια μεταφορά από τις ανθρώπινες επιστήμες, από τις επιστήμες του ανθρώπου, ιατρική, από τέτοιες προπαρασκευαστικές θράσεις και πειρατικά, πειραματικά προγράμματα όλο αντλεί κονδύλη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που μας δυσαρεστεί. Επίσης ένα μεγάλο ποσό αφαιρέθηκε από την υποστήριξη στο πρωτόκολλο της ζάχαρης. Δίνουμε τα χρήματα στις ε, ζαχαροπαραγωγές χώρες, γιατί έχασαν τις ποσοστώσεις τους με την απελευθέρωση του καθεστώτος και έχουμε ένα παρόγραμμα, παρόμοιο πρόγραμμα, απλώς τα χρήματα από, τα, από τη ζάχαρη τα μεταφέρουμε στις μπανάνες. Γιατί δεν δαπανήθηκαν αυτά τα κονδύλια. Συμφωνώ με τη θέση του εισηγητού, αλλά ερώτω, τι έγινε με τα κονδύλια της, μπανάνα, της ε, ζάχαρης. Ευχαριστώ. Ναι, θα πρέπει να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, που πήγαν τα λεφτά της ζάχαρης. Ο κύριος Μπόκρος, νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ακόμη πιο βαθύ. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε ο Ήβο, ότι ο ΠΟΕ αποφάσισε ξεκάθαρα ότι τέτοιου είδους ενίσχυση που αρχικά βοηθούσε τις χώρες ΑΚΕ, που ήταν πρώην βρετανικές ε, και γαλλικές απικίες όλος τυχαίως, όχι ισπανικές, γιατί ο σημερινό δεν επωφελείται. Μερικέ χώρε μόνο επωφελούνταν από την ρύθμιση αυτή. Οπότε το θέμα δεν είναι να γίνει μια ανακύκλωση των κονδυλίων και μια ανακατανομή με διαφορετικό τρόπο. Να πούμε να σταματήσει αυτό το καθεστώς άσχετα με το προϊόν, μπανάνα ή άλλο, και αν μια χώρα χρειάζεται ενίσχυση να το αποφασίσουμε επί τούτου, σε εξατομικευμένη βάση. Και να υποστηρίξουμε συγκεκριμένη περίπτωση άσχετα με το προϊόν. Αν είναι ρύζι, μπανάνα ή ζάχαρη δεν μας ενδιαφέρει. Να δούμε ποιο είδος χρηματοδότησης θα χρησιμοποιήσουμε, το υπαριθμό ένα ζητούμενο και το δεύτερο να είμαστε απόλυτα συμβατοί με τη θέση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου. Ναι, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη συμφωνία που έγινε. Δεν μπορούμε να αφισβητούμε τις λεπτομέρειες. Ή θα τη δεχτούμε ολόκληρη ή θα την απορρίψουμε. Ούτε να για το θέμα αυτό σε άλλε επιτροπές. Ε, Σας ευχαριστώ. αν ξαναπώ τα ίδια με αυτά που λέχθηκαν πριν, ζητώ συγγνώμη. Είχα πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών για να παρουσιάσει μια έκθεση. Όπως είπατε, η συμφωνία είναι take it or leave it. Δύο, μάλιστα, συμφωνίες. Η εμπορική συμφωνία που οδηγεί σε τέλος μια συγκουσιακή κατάσταση και που κανονικά θα έπρεπε να είχε ρυθμιστεί μπροστά στο Διεθνικό Δικαστήριο του ΠΟΕ και εκεί υπάρχουν δύο θέσεις, είτε δηλαδή ε, ένα συμβιβασμός, πιο εύλογο μου φαίνεται αυτό, ή παραμένουμε σε μια κατάσταση σύγκρουσης και την πολιτική την ασκεί τότε το δικαστήριο αντί ημών, αντί των πολιτικών δηλαδή. Η πρώτη υπόθεση είναι η καλύτερη. Για την ίδια τη συμφωνία, η μείωση των ε, δασμολογίων εισαγωγής μπανανών μη ακέ επηρεάζει την κατάσταση των παραγωγών ακέ 40 ευρώ τον τόνο για την εισαγωγή μπανανών ε, λατινοαμερικανικής παραγωγής. Ο πρόεδρος, με συγχωρείτε, μας τα έχει πει αυτά ήδη ο εισηγητής. Αν μπορείτε να συνοψίσετε, ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος, αν μπορείτε να συνοψίσετε το πώς βλέπετε το πράγμα. Ναι, με δύο λόγια, έχετε δίκιο κύριε πρόεδρε. Είμαι εισηγητής για το DCI, Development Cooperation Instrument, που ε, αναφέρεται στην αντιστάθμιση που δίνονται στις χώρες οι οποίες πλήττονται, θίγονται από την Νέα Συμφωνία. Πρόκειται για 190 εκατομμύρια. Η Κομισιόν θα ε, προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας με κάθε μια χώρα ξεχωριστά, αν, επειδή και επειδή η δυνατότητα απορρόφησής τους δεν είναι η ίδια, είτε θα ε, γίνει μια συμφωνία ενίσχυση του προϋπολογισμού τους, είτε ε, του συνολικού είτε κατά τομεί, είτε θα δοθούν τα χρήματα αυτά Δηλαδή θα γίνουν ε, οι δαπάνες αυτές ε, μέσα στα πλαίσια ε, κατασκευής κάποιων έργων ή διεξαγωγή κάποιων προγραμμάτων. Από αυτού κάναμε κάποιες παρατηρήσεις. Ζητήσαμε πρώτα να γίνει μια μελέτη σχετικά με το δρομολόγιο που ακολουθεί η μπανάνα. Θέλαμε να μάθουμε δηλαδή ποιο παίρνει τι λεφτά από το στάδιο της παραγωγής μέχρι το τελικό, την τελική κατανάλωση. Και είδαμε κάτι αρκετά αποκαλυπτικό. Ο παραγωγός στις χώρες ΑΚΕ λαμβάνουν εν τέλει 1,5% της τιμής που πληρώνει τελικά ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Πέραν του δημοσιονομικού δηλαδή, ότι δίνουμε 190 εκατομμύρια. Πρέπει να δούμε και λιγάκι πώς κατανέμεται το ποσό αυτό τα χρήματα αυτά μέσα στην παραγωγή στο εμπόριο της μπανάνας. Γι' αυτό προτιμήσαμε να γίνει μια συζήτηση μέσα στον ίδιο το, τομέα της μπανάνας για να δούμε, χωρίς επιβάρυνση του κοινωτικού προϋπολογισμού, πώς μπορούν να, δοθούν κάποια, να, γίνουν, να ληφθούν κάποια μέτρα λοιπόν, αντιστάθμισης υπέρ των παραγών της μπανάνας. Άλλο σημαντικό είναι να ληφθεί υπόψη μια ιστορική περίοδος στην οποία βασίζονται οι αντισταθμίσεις που να μην είναι πάρα πολύ μακρά, να είναι αρκετά λοιπόν προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα και εν τέλει εμείς ε, έχουμε και εμείς την δική σας ε, ε, επιθυμία να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα γιατί θέλουμε να παραχθούν αποτελέσματα. Οι θυγόμενε χώρες αναμένουν μια απάντηση σύντομα από εμάς Εμεί βέβαια υπεραμεινόμεθα των δικαιωμάτων μας κυρίω για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του, του προπολογισμού. Αλλά θέλουμε βέβαια και να ικανοποιηθούν οι χώρες ΑΚΕ. Αυτά ε, λοιπόν ως ε, πλέον στοιχειώδεις παρατηρήσει. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος αγορητή που έχει εγγραφεί είναι ο κ. Σούριαν. Εγώ νομίζω κύριε Πρόεδρε, βρισκόμαστε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και το βασικό μας θέμα είναι να βρούμε μια λύση σε ένα πρόβλημα. Το ό,τι κάναμε μέχρι τώρα ήταν να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Κανένας δεν μπορεί να θεωρήσει ότι εν τέλει θα κληθούμε να, χρηματο, να χρηματοδοτήσουμε ολόκληρο το θέμα αυτό από το ε, εργαλείο, από το μηχανισμό ευκαμψίας. Δεν μπορώ να πω το 100%. Αυτά είναι ανοησίε του Συμβουλίου που είπε μηδέν από το Flexibility Instrument. Η αρχική πρόταση τη Επιτροπής ε, ήταν ανάμεσα. Όπως είπε όμω η Άννη προηγουμένως σωστά, φύγουν όμως κονδύλια τα οποία και εμά είναι απαράδεκτο να φύγουν. Ε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι... Τι μπορούμε να κάνουμε μάλλον. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία υποτίθεται γινόταν χωρίς πρώτερη ενημέρωση τη αρχή του προπολογισμού. Αυτό όμως αποτελεί πρόβλημα που θα πρέπει να λυθεί μακροπρόθεσμα. Να μην επαναλαμβάνεται δηλαδή. συνηθίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να ξεκινά πράγματα χωρίς να έχει ένα στέρεο ε, δημοσιονομικό υπόβαθρο. Αυτό όμως είναι απαράδεκτο. Βρισκόμαστε λοιπόν στην φάση τώρα όπου ακούγονται διάφορα. Να προχωρήσουμε τώρα λίγο και να γίνει αυτό ελπίζω να είναι εδώ παρούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να με ακούει εάν προτείνουν κάτι που είπε και ο Επίτροπος στη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου και εγώ ήμουν τότε αντίθετος και όφιλα να είμαι και αντίθετος διότι αυτή ήταν η βασική αρχή είτε συμφωνούμε με όλα είτε με τίποτα. Ο κύριος Λεβαντόφσκι λοιπόν πρότεινε ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με το μέρος εκείνο του redeployment όπου δεν ε, σημαίνει κάποιες δαπάνες και δεν συνεπάγεται δηλαδή δαπάνες στη διάρκεια του τριμερού διαλόγου, εγώ δεν είχα την εντολή να το αποδεχτώ αυτό. Αν όμως δεν υπάρχει περιθώριο ελιγμών τους επόμενους μήνες, νομίζω ότι μπορούμε να δεχτούμε μια ενδιάμεση λύση. Όχι για το σύνολο των 75 εκατομμυρίων, αλλά για ένα εύλογο μέρος του ποσού αυτού, που να μην αποβεί ιδιαίτερα οδυνηρό. Εάν η Επιτροπή μας δεχθεί την προσέγγιση αυτή, αυτό θα είναι ένα μήνυμα καλής θέλησης. Λοιπόν, λέμε απλώς καλά λόγια, αλλά στην πραγματικότητα είναι, έχουν σταματήσει τα πράγματα τώρα. έχοντας μια επαρκή πρόταση, εγώ ως εισηγητής από την πλευρά του προπολογισμού, δεν θα είμαι αντίθετος. Ταυτόχρονα προωθείται το θέμα της νομικής βάσης και αυτό πάλι είναι εκδήλωση της καλής θέλησης του Κοινοβουλίου, ότι θα, θέλουμε, θα θέλαμε να γίνει δηλαδή, αλλά είναι πάρα πολύ περίεργο και πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι. Πώς είναι δυνατόν να γίνει διεθνή συμφωνία χωρίς ε, νομική βάση. κάτι τέτοια καταστρέφουν την αξιοπιστία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να συνάπτει ε, διεθνείς συμφωνίες και μετά να ανακαλύπτει ότι έχει δυσκολία να πληρώσει. Ε, πρέπει να λυθεί αυτή η κατάσταση. Αν είμαι καλά πληροφορημένος, αυτά τα 75 εκατομμύρια αποτελούν τμήμα της συμφωνίας που περιλαμβάνει αυτή την ανάλυση των ποσών, εάν στο τέλος δεν μπορούμε να δώσουμε τα χρήματα, τότε παραβιάζει τη συμφωνία. Ποιος ευθύνεται. Είμαι βέβαιος ότι δεν ευθύνεται η Επιτροπή Προϋπολογισμών για τη δημιουργία αυτής της κατάστασης. Αλλά η ευελιξία μας συνδέεται με το μηχανισμό ευελιξίας και εν μέρη μπορούμε να είμαστε και ευέλικτοι εάν δεν θυγούν τα κονδύλια εκείνα τα οποία ε, έχουν πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Θα μπορέσω λοιπόν να δείξω κάπως περισσότερη ευελιξία ή ευκαμψία για να προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει δεκτή αυτή η θέση του Συμβουλίου. Και θα χρειαστώ την υποστήριξή σας για να φανούμε όλοι ε, αμετακίνητη το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο άλλος εισηγητής, ευχαριστώ μάλλον εσάς κύριε άλλη εισηγητά, ακούσαμε όλοι και όσοι εκπροσωπούν άλλα θεσμικά όργανα εδώ, τα όσα είπατε. Ας μείνουμε σε αυτά, για αυτό το σημαντικό θέμα. Έχετε λοιπόν λάβει υπόψη τις, ε, τα γραπτά κείμενα και τις θέσεις των συγητών. 15 Ιουλίου μεσημέρι η προθεσμία κατά τροπολογιών και έγκριση τον Σεπτέμβριο υπό την επιφύλαξη των όσων θα συμβούν μέχρι τότε και εφόσον όσα προτείνει ο συγητής και όπως υπενθύμησε ο Λάσλο Σούριαν για τα όσα είπε ο Επίτροπος Προϋπολογισμών στον τριμερή διάλογο ενδεχομένω να δούμε άλλη, άλλη, άλλη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να μας επιτρέψει να εργαστούμε σε πιο ξεκάθαρες βάσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Σιγητά. Το αποκορύφωμα τώρα των εργασιών μας. Ο Ράιμερ Μπέγκε, η αποθέωση. Ο Ράιμερ Μπέγκε πριν να πάμε στις θερινές διακοπές, ο οποίος θα μας παρουσιάσει όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουμε αφήσει για το τέλος. Και αυτή τη συζήτηση αμέσως πριν να ε, συναντήσουμε τον Υφυπουργό Βάτλι στους συντονιστές. Τα διάφορα θέματα, midterm review, το παγκόσμιο της αγώνας, ε, το μέλλον του ε, κοινοτικού προϋπολογισμού και το καθεξής. Ωραία äh, Θα είμαι σύντομος σήμερα κύριε Πρόεδρε, αφού δεν πρόκειται για τίποτε άλλο για, παρά για το follow-up μιας διαδικασίας που έχει συμφωνηθεί εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στη βάση των συζητήσεων και ερωτήσεων που έχουν γίνει προς τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με την midterm review που τη συζήτηση κάναμε ήδη τον Ιούνιο στο Στρασβούργο. Έχετε μπροστά σας ένα σχέδιο για μια λεγόμενη έκθεση interim Ομολογώ ότι αρχικά ήθελα να διαβάσω την έκθεση σε όλους την Παρασκευή, αλλά καμιά φορά, όπως συμβαίνει καμιά φορά στο κοινοβούλιο, με εμπόδισε το λεγόμενο tabling office. Σύμφωνα με το άρθρο 81 παραγράφος 3 υπάρχουν ορισμένα φορμά μέσα στα οποία πρέπει να χωρέσει μια έκθεση. Εξεπλάγει για τη διαδικασία αυτή. Είχα την ευκαιρία βέβαια ευτυχώς να συζητήσω με άλλους συναδέλφους για τις απόψεις των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Άκουσα άλλωστε και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Έτσι, σε επίγουσα διαδικασία χρειάστηκε να προσαρμόσω κάπως τα πράγματα και βέβαια να φροντίσω να δω και όλας ώστε με αυτή την ανάγκη να υπαχθεί σε αυτό το συγκεκριμένο διοικητικό φορμά ε, η έκθεσή μου τελικά να ε, χάσει λίγο το χαρακτήρα της. Δεν προλάβαμε με λίγα λόγια τις προθεσμίες. Δεν μου αρέσει να με βάζουν σε τέτοια διοικητικά στενά, ας πούμε έτσι, σε αυτό το φόρμα. Αυτά θα πρέπει να συζητηθούν και στην διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών. Σχετικά δηλαδή με το τι μορφή πρέπει και καλά να λάβει μια έκθεση. Ένα συζητήτη ο οποίος έχει διαμορφώσει μια έκθεση σε βάση μιας ε, διάρθρωσης που έχει σκεφτεί, ξαφνικά βλέπει ότι την ανατρέπουν. Δεν μου αρέσει λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο κινείται η διαδικασία. Μια πρόοδο ότι στο μέλλον το tabling office θα ενταχθεί στις ε, γραμματείες των επιτροπών και άρα στο μέλλον θα υπάρξουν κάποιες ε, πιο θετικές συνέργειες, ας το πω έτσι, και οι δυνατότητες συνεργασίας θα είναι ε, βελτιωμένες. Αυτά ως μια πρώτη προκατακτική παρατήρηση, διότι όπως είπα εξεπλάγει από αυτό που είδα να βγαίνει από το tabling office μετά από ό,τι θα τους είχα τροφοδοτήσει εγώ. Πράγματι, στην βάση της σημερινής συζητήσεως έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε τροπολογίες μέχρι τις 21 Εβδόμου και να γίνει η ψηφοφορία μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου. Αναμένοντας το τι θα πράξει το Συμβούλιο, εάν δηλαδή θα τα καταφέρουμε με την Βελγική Προεδρία να διεξαγάγουμε εντατικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, είτε εάν η πλευρά του Συμβουλίου δεν είναι διατεθειμένη να διδαχθεί αρκετά από τη διαδικασία SWIFT. Γιατί βέβαια υπάρχει διαθεσμική συμφωνία η οποία πρέπει να προσαρμοστεί στην βάση της συνθήκης της Λισαβόνα. Πρόκειται για πολιτική συμφωνία όμως η οποία μπορεί να επιβιώσει και να προσαρμοστεί μόνο με συμφωνία όλων των μερών. Και αυτή η προσαρμογή πρέπει να έχει και ένα πολιτικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να είναι μοναχά τεχνική και χρειάζεται επομένως και την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που να εκφράζεται με ειδική πλειοψηφία. Είναι λοιπόν σωστό να ακολουθηθεί αυτή η οδός μιας ενδιάμεσης έκθεσης, αφού δεν υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση. Στην διατύπωση αυτής της ενδιάμεσης έκθεσης, μία από τις κατευθυντήριες ας πούμε σκέψεις μου, ήταν να δοθούν ξεκάθαρα σύντομα μηνύματα προς Κομισιόν και Συμβούλιο και σε ένα παραπέρα βήμα, αρχάς Σεπτεμβρίου, να συντάξω ένα έγγραφο εργασίας και στην βάση και των συζητήσεων που θα γίνουν εδώ στην Επιτροπή, και να εμπλουτιστούν οι συζητήσεις και με τροπολογίες για την περαιτέρω διαμόρφωση του προπολογισμού τα επόμενα χρόνια. Αναμένω τροποποίηση των προτάσεων της Κομισιόν μετά και από τις επικείμενες συζητήσεις που θα γίνουν με το Συμβούλιο. Η παράκτησή μου λοιπόν είναι να μην προχωρήσουμε σε υπερβολικά σε υπερβολικά λεπτομερείς διευκρινήσεις. Δηλαδή για το ποια θα είναι τα κονδύλια συγκεκριμένα για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων ή για τον μηχανισμό ευκαμψίας. Για τα ποια πράγματα πρέπει να επιτύχουμε μέχρι το 2013 σε ό,τι αφορά τα διαθέσιμα περιθώρια λιγμών ή τι μπορεί να κοστίσει για παράδειγμα η δημιουργία αποθεματικών σε σχέση με το 0,03% του ΑΕΠ. Και επειδή σύμφωνα με τις νομικές υπηρεσίες δεν θα είναι δυνατόν πλέον η διαθεσμική συμφωνία να τροποποιηθεί, θα πρέπει αυτά να γίνουν σαφή με τροπολογίες δηλαδή προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ακόμα όμως αυτό είναι πρόωρο. Και αυτά που συζητήθηκαν στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπου δηλαδή αναφερθήκαμε στην απλούστευση της διαδικασίας και άλλων δημοσιονομικών διαδικασιών, τα είπαν προηγουμένως Κάλφιν και, και ε, Σούριαν, τι κάνει ακριβώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ασκεί πίεση στην αρχή του προπολογισμού, ώστε να λάβει κάποιες αποφάσεις για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα στο μέλλον θα πρέπει η διαθεσμική συμφωνία να γίνει αντικείμενο επανεπεξεργασίας ώστε στο μέλλον να μην υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση των μεν από τους δε, όπως έπραξε η Κομισιόν τους τελευταίους μήνες απέναντί μας. Αυτά πρέπει να εγγραφούν στη νέα διαθεσμική συμφωνία, ώστε στο μέλλον η ε, συνεργασία να γίνεται σε μια διαφορετική βάση. Στο κείμενό μου περιορίζομαι ιδίω στο να καταστήσω για άλλη μια φορά σαφές στις επιμέρους παραγράφους ότι θεωρώ απαραίτητο εν ώψη των νέων προκλήσεων και της καταστάσεως της ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής και παρόλη την ε, υφιστάμενη κατάσταση ότι είναι ε, απαραίτητο να γίνει, απαραίτητο να γίνει πιο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες μεταξύ των θεσμικών οργανών. ότι Εμείς περιμένουμε να κάνουν περισσότερα Επιτροπή και Συμβούλιο και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να έχει στη διαθεσή της επαρκή κονδύλια και εδώ τονίζω επίσης ότι δεν είναι δυνατόν ούτε παραδεκτό ως εναλλακτική επιλογή μια δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες μέλη να τίνουν μέσω άλλων μηχανισμών, είτε μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είτε μέσω κρατικών εισφορών, είτε με άλλες δραστηριότητες, να υποσκάπτουν την κοινωτική μέθοδο του προϋπολογισμού. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα συγκεκριμένο προβληματισμό και πρέπει να συζητηθεί και στις διαπραγματεύσεις τώρα, αλλά και σε επιμέρους project που θα ε, γίνουν στο μέλλον αλλά και στην επόμενη, στον επόμενο πολιετή δημοσιονομικό σχεδιασμό. Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό πρόβλημα ή και πρόκληση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τοποθετηθούμε και για αυτά. Στο κείμενο διασαφίζω για μια φορά ακόμη ποια είναι η κατάσταση από άποψη κανονισμού, για ποιο λόγο χρειαζόμαστε αυτή την και πολιτική προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τονίζω και πάλι ότι το Κοινοβούλιο δεν θα μπορέσει να αποφύγει να τοποθετηθεί ε, απέναντι στις θετικές και αρνητικές προτεραιότητες του προϋπολογισμού και τονίζω και πάλι με έμφαση ότι οι νέες δημοσιονομικές προκλήσεις δεν θα μπορέσουν πλέον να αντιμετωπιστούν με απλές μετακινήσεις ε, κονδυλίων ή με απλούς μηχανισμούς που και ότι επομένω θα χρειαστούν και από την πλευρά του Συμβουλίου και από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νέες προτάσεις πώς θα μπορέσει να εξεταστεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός μακροπρόθεσμα και σε συνδυασμό με του εθνικού προπολογισμού, Τι σημαίνει αυτό άλλωστε για το εθνικό και για το περιφερειακό επίπεδο. Τα πράγματα αυτά τα διαλαμβάνω στο κείμενο και αναφέρομαι επίση και στην επανεξέταση του προπολογισμού που προβλέπεται για τον Σεπτέμβριο και για τι αντιφατικέ ε, συμπεριφορέ ε, τη Επιτροπή και του Συμβουλίου είτε πρόκειται για την συμφωνία για την μπανάνα, είτε πρόκειται για άλλες συζητήσεις οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν. Αναμένουμε επίσης η συνολική αυτή συζήτηση για τις νέες αυτές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων κλπ. Αυτά πρέπει να υπαχθούν σε τη συζήτηση αυτή. Ή αλλιώς θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μακροσκελείς και δύσκολες διαδικασίες του προπολογισμού και το Συμβούλιο και η Επιτροπή οφείλουν να αντιληφθούν ότι μια θετική συνεργασία είναι προς όφελος όλων. Το θέμα επίσης της ευκαμψίας και των περιθωρίων τίθεται επίσης στο κείμενο. Εδώ πρέπει να συζητήσουμε λίγο και να στοχαστούμε στη διάρκεια των θερινών διακοπών πώς εν ώψη αυτής της δύσκολης κατάστασης της ευκαμψίας ή της αναθεώρησης κάτω από το 0,03% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, πώς θα βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε το περιθώριο αυτό ήδη από την αρχή των διαπραγματεύσεων και να μην δεχθούμε απώλεια ευκαμψίας και ήδη από την αρχή των διαπραγματεύσεων να βρεθεί μια διέξοδος μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Εξαρτάται βέβαια από ποια διέξοδο θα βρεθεί. Αυτό θα έχει όμως κάποια συνέπεια για το ποιου μηχανισμούς ευκαμψίας χρειαζόμαστε ώστε να εξασφαλιστεί αυτό το απόλυτο ελάχιστο. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα δηλαδή αυτό που θα έχουμε για ειδικά αυτό το τμήμα του 0,3% του 0,03%. Το θέμα του του προπολογισμού επίσης τίθεται και εν τέλει πάλι περιλαμβάνεται μια παράγραφος που ασχολείται με αυτήν την δέσμη του μηχανισμού σταθερότητας και πράγματα που συζητήσαμε και πριν, ότι δηλαδή εάν θεωρήσουμε ότι ο μηχανισμός αυτός πρέπει να αποδίδει και οι εγγυήσεις και ε, ε, ε, εφόσον δηλαδή κληθεί ο μηχανισμός σταθεροποίησης και οι σχετικές ρυθμίσεις να λειτουργήσουν, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική συνεργασία, βεβαίως με διαφάνεια, μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το Κοινοβούλιο δείχνει, με το, στο παράδειγμα αυτό, ότι λειτουργεί με απόλυτα υπεύθυνο τρόπο και ότι αναμένουμε περισσότερο υπεύθυνο τρόπο και από τα άλλα θεσμικά όργανα στην αντιμετώπιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα παρακαλέσω οι πολιτικές ομάδες να εξετάσουν προσεκτικά το κείμενο, να διατυπώσουν τροπολογίες και θα έχουμε χρόνο πριν από την ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο στην Επιτροπή να εγκύψουμε στις διάφορες λεπτομέρειες οι οποίες ενδεχομένως θα είναι απαραίτητο να συζητηθούν, να συνεννοηθούμε, να δούμε και αυτές τις τάσεις να δούμε πού πρέπει να υποβάλουμε πολύ συγκεκριμένες τροπολογίες για την τροποποίηση της Διαθεσμικής Συμφωνίας και να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία, όπως είπα, σταδιακή. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Merci, cher très, très Σας ευχαριστούμε, κύριε Σιγητά. Ήσασταν σαφέστατος. Και πολύ σοφό αυτό το διάβημα. Και μάλιστα είναι σαφές ότι αν σήμερα δεν είχαμε αυτή τη μόνιμη πίεση του Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα της δικής μας Επιτροπής, δεν θα είχαμε καν διάμεση αναθεώρηση. Και πραγματικά είναι καταπληκτικό ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το Συμβούλιο ε, ζήτησε και εμείς ε, ασθενιστήκαμε αυτή την έτσι και, την, και υπερθεματίσαμε, να ε, επεκταθεί αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση και στην απόφαση δημοσιονομικών προοπτικών του Συμβουλίου 2007-2013 και να καλύπτει και τους ιδίους πόρους, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της και να καλύψει και κάποιες πολιτικές όπως την κοινή γεωργική πολιτική. Αυτό το ζήτησαν οι Βρετανοί. Οπότε είναι περιεκτική αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση η εμβέλειά τη είναι ευρεία. Και αυτό φαίνεται το Συμβούλιο ξαφνικά να το, ξε... να, έχει... να το έχει ξεχάσει. Και αυτό που είναι ακόμη πιο περίεργο είναι ότι φαίνεται να το έχει ξεχάσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάθε φορά που λέμε κάτι τέτοιο, ε, είναι σαν να τους ε, βρίζουμε, σαν να τους προσβάλλουμε. Άνω ποταμών. Ενώ υπάρχουν ένα σωρό άλλοι λόγοι που δεν υπήρχαν καν το 2006 πολύ περισσότερα επιχειρήματα σήμερα που συνηγορούν υπέρ της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Για παράδειγμα, το μείζον επιχείρημα είναι η θέση ισχύ τη ε, συνθήκη Λισαβόνα με τι νέε αρμοδιότητε. Τότε το 2006 δεν είχαμε συνθήκη τη Λισαβόνα, είχε απορριφθεί η συνταγματική συνθήκη. Δεν είχαμε καν την ελπίδα ότι θα εγκρινόταν η δεύτερη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και έχουμε φυσικά και την οικονομική κρίση, την τελευταία διεύρυνση του 2007. Ο κύριος Κάρφιν τότε, το 2006, δεν ήταν καν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Κάρφιν θέλει τα λεφτά του πίσω, όχι πίσω μάλλον, θέλει το μερίδιό του. Διεκδικεί το δίκαιο μερίδιό του. Κι αν δεν ασκούσαμε εμείς την πολιτική πίεση που θέλουμε να κρατήσουμε μέχρι τελευταία σαρανίδος, μέχρι το Σεπτέμβριο, θα είχαμε δύο πολύ ισονοσημασίες ε, σχέδια ε, ενδιάμεση αναθεώρηση των προοπτικών για ένα-δύο προγράμματα που είναι προσφυλίτε στην Επιτροπή της στο Συμβούλιο. Δεν είναι σωστό αυτό, δεν είναι ορθός τρόπος μεθοδολογίας. Το είπαμε προς και κατευθύνσεις με κάθε δυνατό τρόπο και δημόσια και ιδιωτικά και συνεχίζουμε να το διατρανώνουμε όσο πιο χειρά μπορούμε και μέσω αυτής της έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Ενδιάμεση έκθεση στα πλαίσια της διαδικασίας» και που δίνει συνέχεια στις προηγούμενες προφορικές ερωτήσεις. Και σας υπενθυμίζω το χρονοδιάγραμμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν τις προτάσεις και μάλιστα ακόμη και το, από το Σεπτέμβριο. Οπότε στις 21 Ιουλίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση Μπέγκε. Ακούσατε τις προτάσεις του εισηγητού. 21 Ιουλίου σας έμειναν λίγες μέρες ακόμη, ώστε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 13 Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια, στη δεύτερη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Έχουμε ακόμη 20 λεπτά περίπου. Θα ακούσουμε μερικούς ομιλητές. Η κυρία Γιάνσεν. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ το Ράιμερ για την ιόβια υπομονή του και την επιμονή του που έδειξε στο θέμα αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνουμε κάτι και παρελειμμένος μάλιστα και έχουμε συγγυηθεί και από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαν ε, ε, να μιλάμε σε κουφού. Φωνή βόντω ότι ερήμο, σαν να παίζουμε ένα τείχο. Χτυπάμε τον τείχο και τον μπαλάκι επιστρέφει. Συμφωνώ με το κείμενο, παρόλο που ήταν πολύ μετριόφρον και ταπεινόφρον ο, ο Ράιμερ για το περιεχόμενο. Πιστεύω πάντως ότι το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει πλήρω τη συζήτηση που είχαμε επ' ευκαιρία των προφορικών ερωτήσεων, αλλά και προηγούμενες συζητήσεις και αντανακλά την απογοήτευσή μας και τη ματέωση που αισθανόμαστε και μάλιστα μια σημαντική απογοήτευση αφορά το θέμα το πρόγραμμα ΙΤΕ για την ενέργεια από τη σύνδεξη. Ένα θέμα που το εξετάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το Συμβούλιο τώρα βρήκε μια λύση που λέει ότι το 2012 και 2013 θα χρηματοδοτήσουμε το 1,4 δις με την περικοπή άλλων σχεδίων από το 7ο ερευνητικό πρόγραμμα πλαίσιο. Αν το συζητούσαμε, ίσως θα μπορούσαμε φέτος ε, ή άλλες χρονιές στο παρελθόν να διαπιστώνουμε ότι υπήρχε υποαπορρόφηση σε κάποια προγράμματα. Αλλά δεν υπάρχει ένδειξη για κάτι τέτοιο. Οπότε, έχετε μια σημαντική προτεραιότητα στη στρατηγική του 2020. Μια ύψη προτεραιότητα που την έχουν αστερνιστεί και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και αυτή την προτεραιότητα τη συρρυκνώνουμε προς όφελος μιας άλλης που είναι ίσονος σημασίας και αβέβαιης έκβασης. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Και ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι αντί να έρθει το Συμβούλιο και να μας πει ε, με το σωστό τρόπο μήπως μπορούμε να βρούμε καμιά λύση, ασκεί αφόρητη πίεση προσωπικά στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό που δεν βρέθηκε η σωστή διάβλος για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων από την Επιτροπή. Και δυστυχώς φαίνεται δεν άκουσε η Επιτροπή αυτά που είπαμε στον κύριο Λεβαντόφσκι για αυτό που του ζητήσαμε όταν συμφωνήσαμε, όταν δώσαμε το πράσινο φως για το διορισμό του στη θέση του Επιτρόπου. Μέχρι τώρα θα πρέπει ήδη να είχαμε την πρόταση για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Που θα ήταν χρήσιμη όχι για μας, αλλά πρώτα απ' όλα θα ήταν ωφέλιμη για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να ελέγξει τα περιθώρια ελαστικότητας και τις δυνατότητες των τελευταίων χρόνων των δημοσιονομικών προοπτικών. Είναι σαν να πιστεύουν όλοι ότι μας νοιάζει μόνο να υπερβούμε τα ανώτατα όρια. Αντιλαμβανόμαστε τη δινή οικονομική κατάσταση των κρατών μελών και θέλουμε να εξετάσουμε λεπτομεριακά τα προγράμματα, να δούμε πού υπάρχει υποαπορρόφηση, που υπάρχουν δυσλειτουργίες, ώστε να καταρτήσουμε ένα πιο σωστό και σταθμισμένο κατάλογο προτεραιοτήτων, αλλά να βρούμε μία λύση, αντί να έχουμε αποσπασματικές προτάσεις και να κόβουμε από εδώ και να ράβουμε από εκεί, χωρίς να έχουμε τη γενική εικόνα της κατάστασης. Ελπίζω να το λάβει αυτό υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην κοφεύσει αλλά πραγματικά μας είναι απαραίτητη πια η ενδιάμεση αναθεώρηση. Και θα πρέπει να δώσει μια απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είναι αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση. Αυτό είχε υποσχεθεί ο κ. Λεβαντόφσκι ότι θα μα τη στείλει μετά το διορισμό του. Και πραγματικά είναι εξοργιστικό που ακόμη την περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε, Αν, γιατί πραγματικά μας θύμισες ότι όταν ε, ο φίλος μας ε, Λεβαντόφκη πέστη την ακρόασή μας ε, είχε αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή, θα ήθελα να κάνω μια διόρθωση όσον αφορά την προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Είναι 22 και όχι 21 Ιουλίου, γιατί 21 Ιουλίου ε, είναι η ημέρα της εθνικής γιορτής ε, του ε, Βελγίου. Θα έχετε διαπιστώσει όλοι ότι έχουν ξεκινήσει να βάζουν εξέδρες μπροστά από το βασιλικό παλάτι κτλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σίγουρα θα πρέπει να κρατήσουμε αμύωτη την πίεση, γιατί τα αιτήματά μας είναι σοβαρά, θεμελιωμένα, τεκμηριωμένα και έχουν και νομική βάση. Έχουμε μια στρατηγική, ξεκινήσαμε με την προφορική ερώτηση, η συνέχεια δίδεται με την ενδιάμεση αυτή έκθεση και θα συνεχίσουμε μέχρι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Και ευτυχώ υπάρχει η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να δείξουμε τη δύναμή μα απέναντι στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μπέγκη γιατί μα επέτρεψε να εμπλακούμε ενεργά στην εκπόνηση του σχεδίου έκθεσης και επίση για την καλοσύνη να συμπεριλάβει σχεδόν όλες τις προτάσεις ε, που καταθέσαμε. Ζητώντας το ακριβώ να τις συμπεριλάβει. Γενικώ συμφωνούμε σε αδρές γραμμές. Ε, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες. Θα εξετάσουμε πιο διεξοδικά την τελευταία πρότασή του και θα υποβάλουμε αντίστοιχα τροπολογίες. Συμφωνώ μαζί σας ότι η έκθεσή μας θα πρέπει να είναι απλή, σαφής και όχι υπερφορτωμένη με λεπτομέρειες για να είναι ξεκάθαρη φως φανάρι θέση μας. Το θέμα της ελαστικότητας πάντως θα πρέπει να αναφέρεται με τη δέουσα σημασία γιατί είναι ζωτικό για οποιοδήποτε δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κέριο ζήτημα η ελαστικότητα. Οπότε θα πρέπει η έκθεση αυτή όχι μόνο να προτάσει τη θέση μας και να απορρίπτει τη θέση του Συμβουλίου για το βαθμό ελαστικότητας του δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον μία πρόταση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε ό,τι αφορά το βαθμό ελαστικότητας ε, που διεκδικούμε για να μάθουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή ποιε είναι οι προθέσεις μας. Πάντως ε, υπάρχει σύμπνοια και στόχος μας είναι να εγκρίνουμε την έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία για να δείξουμε την ε, δύναμη, την πυγμή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Έλγα Τρυπέλ είναι η τελευταία μιλήτρια. Διαπιστώνω ότι ο εισηγητής μας κυρίως στα γυναικεία πνεύματα εξάπτει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον Ράιμερ για την σύνταξη της έκθεσής του. Όταν ήρθα να γίνω Ευρωβουλευτής και ζήτησα να ε, ενταχθώ εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό που θα αντιμετωπίζουμε συχνά και ξανά και ξανά είναι αυτό το, είναι αυτός ο διαθεσμικός αντάθετο πόλεμος. Αυτά όλα είναι εξαιρετικά εξοργιστικά. Και αν σκεφτεί κανείς και τι σημαίνει αυτό και προς τα έξω για την αποδοχή από πλευρά των πολιτών. Βρίσκω ότι η ζημιά είναι μεγάλη εκεί. Εξεπλάγιν τα πράγματα είναι πραγματικά τόσο άσχημα. Δεν το περίμενα. Αναμένει κανείς εντιμότητα στις σχέσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Το δεύτερο πρόβλημα, που σωστά το είπε πάλι ο Ράιμερ, Νομίζω ότι πρόκειται για πολιτική αποτυχία. Ας δούμε τις δημοσιονομικές συζητήσεις που κάνουμε και τις διαδικασίες με συζητήσεις και ξανά συζητήσεις επί μήνε με όλες αυτές τις μεταφράσεις όταν μιλούσαμε για το Γαλιλαίο ή για το Recovery Plane. Αυτή η πολιτική της Κομισιόν και του Συμβουλίου που έρχονται και αποφασίζουν καινούργια πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν με την, με την ε, δομή του προπολογισμού. Είναι πολιτικό πρόβλημα, ότι δηλαδή ο προπολογισμό είναι προβολικά άκαμπτος και απερχαιωμένο ώστε δεν αντιμετωπίζονται σωστά ε, οι ανάγκε, Αλλά δεν υπάρχει και η πολιτική δύναμη μέσα από όλα αυτά τα συμπτώματα τα οποία κάθε τόσο αντιμετωπίζουμε με διάφορα μέσα να αποφασίσουμε να προχωρήσουμε σε νέες δομές. Μέχρι τώρα όλα τα φορτώνουμε σε αυτή την περίφημη review που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει. Και όταν έγινε η ακρόαση του Λεβαντόσκη, με διαφορετική ε, στάση στην ψηφοφορία, ήταν σαφές τότε ότι είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες ανάληψης δράσης από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά είχα πει εγώ τότε ότι πρέπει να αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν μπορεί να αρκείται στο ρόλο απλώς ε, του ενός πολιτιολόγου ο οποίος θα μας εξηγεί ποιες είναι οι θεσμικές σχέσεις των οργάνων. Και αυτά τα είπε πάλι ο Ράιμερ, η εξέφραση το παράπονο, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά ισχυρή και επομένως δεν μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη μιας πραγματικής πολιτικής πρωτοβουλίας. Τρίτη παρατήρηση που την ανέφερε και η Ίγκε Γκρέτσλερ. Όντως, κύριε Πρόεδρε, όταν βλέπουμε την τροχοπέδη του ελίματος και του χρέους, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε ό,τι κατεβεί στο κεφάλι μας ε, και ότι θα πρέπει με ευφυή τρόπο να εναρμονιστούμε οι μεν με τους δε και να συνεννοούμαστε. Και νομίζω ότι αυτό καταφέρεται ε, σαφώς σε πολλές παραγράφους του κειμένου του συναδέλφου Μπέγκε. Θα χρειαστεί να θέσουμε νέες προτεραιότητες στη δράση μας έτσι ώστε η όποια κοινοτική ενωσιακή δράση να ε, έχει προστιθέμενη αξία. Πώς είναι δυνατόν επίσης να ε, διασυνδέσουμε με ευφυή τρόπο τους εθνικούς προπολογισμούς με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί διαφορετικά ε, πολιτικά και δημοσιονομικά η όποια προσπάθειά μας θα αποτύχει. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό να πούμε ότι γνωρίζουμε βεβαίως ε, ότι, το, ότι η κατάσταση η οικονομική μπορεί να είναι δυσχερής σε πολλές χώρες μέλη, αλλά ε, ότι από πολιτικής απόψεως θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα, ε, ποια είναι τα διακυβεύματα πραγματικά, γιατί διαφορετικά φοβούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα έχουν κανένα ενδιαφέρον για μας και οι Ευρωπαϊκή Ένωση σαν θεσμός δεν θα παρουσιάζει καμία έλξη. Είναι σημαντικό να ε, ε, δούμε ε, βεβαίως και το θέμα του... Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιηθούν χρήματα. Έχουμε δώσει πολλά χρήματα για αυτό το πρόγραμμα μέσα σε έναν ανεπαρκή προϋπολογισμό. Και αναρωτιέμαι, και φαντάζομαι θα αναρωτηθούν και άλλοι, μα δεν υπάρχουν πιο επίγοντα θέματα. γιατί ε, φοβούμε ότι τελικά θα αφήσουμε πίσω μας ένα τεχνολογικό ερείπιο το οποίο δεν θα λειτουργεί καθόλου. Πρέπει λοιπόν να συντονιστούμε και αυτή τη στιγμή λαμβάνοντας ε, υπόψη ε, τα οικονομικά προβλήματα, την οικονομική δυσχέρεια, ε, πιστεύω ότι δεν είναι η κατάλληλη ώρα για να ξεκινήσουμε προγράμματα τύπου ITER. Δεν λέω ε, να εγκαταλείψουμε όλα τα τεχνολογικά προβλήματα γιατί υπάρχουν ε, προγράμματα συγγνώμη, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία θα την ανταγωνιστικότητά μας ε, στη διεθνή σκηνή. Λέω απλώς ότι θα πρέπει εδώ να πάρουμε και κάποιες πολιτικές αποφάσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα, περισσότερη τεχνολογία αλλά σίγουρα όχι για, έναν, για ένα πρόγραμμα που θα ασχολείται με την τήξη και τα λοιπά. Δεν θα επισέλθουμε στη συζήτηση επί της ουσίας. Πάντως, όπως είπε και ο Ράιμερ, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τη μεγάλη δυσκολία που προέρχεται από την ακαμψία του προϋπολογισμού. Πριν από 25 χρόνια συνήψαμε τις πρώτες διοργανικές συμφωνίες ακριβώς για να χαλαρώσουμε αυτή την ακαμψία του άρθρου 272 τότε, της τότε συνθήκης και με κάποια ανώτατα όρια και υποανόφλια ε, δημιουργήσαμε ένα κλειό ασφυκτικό. Ένα είδος ζωλομανδία που μας φέρνει σε καταστάσεις πολύ δύσκολες. Σχεδόν αδιέξοδες. Και όταν ακούμε πολλές φορές τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τονίζουν το πρόβλημα αυτό της πολιτικής αναγκαιότητας και της συμφωνίας του 2006 να καταρτιστεί μια ενδιάμεση αναθεώρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας απαντά «Μα πώς μπορούμε τώρα να προτείνουμε αύξηση των ανώτατων ορίων δεδομένης της ε, γενικής ε, οικονομικής κρίσης». Το πνεύμα όμω τη ενδιάμεση αναθεώρηση δεν είναι μια συστηματική αύξηση όλων των κεφαλαίων μέχρι το τέλο ε, τη περίοδου των δημοσιονομικών προοπτικών. Στην συγκεκριμένη περίοδο που διανύουμε, θα ήταν λογικό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει αυτή τη στιγμή θέλουμε να ελέγξουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, αλλά δεν θα αυξήσουμε τον κυρωτικό προπολογισμό. Ο προπολογισμό του 2011 θα έχει μηδενική αύξηση, αλλά το 2012 και 2013 θα δώσουμε έμφαση σε κάποιες πολιτικές προτεραιότητες, ε, όπως προκύπτουν από το πρόγραμμα το 2020. Δεν είναι επειδή θα κάνουμε την αναθεώρηση ε, ότι συστηματικά θα τα δαπανούμε περισσότερα, απλώς ε, πιο ορθολογική χρήση των κονδυλίων, καλύτερη χρησιμοποίηση. Αλλά αν η Επιτροπή έχει το μονοπόλιο των νομοθετικών προτάσεων, από τη στιγμή που δεν υποβάλλει τι προτάσει τη, εμεί μένουμε με δεμένα τα χέρια. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντίθετα με αυτά που προέβλεπε η Διοργανική Συμφωνία, ουσιαστικά μα δεσμεύει και μα βάζει φραγμού. Ο Γκέραν Φέρμ ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι Και πάλι θα, θα ήθελα να πω ότι αναπληρώνω τη Γιούτα Χάουγκ εδώ. Έστειλε ένα σημείωμα για, με τις σκέψεις της. Συμφωνώ απόλυτα με την ενημέρωση και την έκθεση του Ράιμερ. Και έχω ένα επιπλέον σχόλιο εκ μέρους της ε, Έχουμε στο 1.6 τον επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων και το κατά πόσο θα πρέπει να ζητήσουμε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλει τέτοιες προτάσεις ανακατανομής και επαναπροσδιορισμού των προτεραιοτήτων. Χθες, τα εξετάσαμε χθε με την κυρία Γεντζεγεύσκα και είπε ξεκάθαρα ότι δεν θα υποβάλει προτάσεις για ανακατανομή και επαναπροσδιορισμό των προτεραιότητων. Θα το συζητήσουμε αν μας υποβληθεί ως πρόταση, αλλά δεν θα αναλάβουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία. Ενώ φαίνεται ότι το κείμενο αυτό ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποβάλει πρόταση ανακατανομή ή επαναπροσδιορισμού. Κάτι που έρχεται σε αντίφαση με αυτά που μα είπε χθε η Σιντόνια στην έκθεσή τη, η κυρία Γιάννη Ζαγεύσκα. Μήπως αυτό το σημείο θα μπορούσε να το διορθώσει ο Ράιμερ, να τροποποιήσει κάπως τη διατύπωση ίσως και να διαγράψει κάποια τμήματα αυτής της παραγράφου. Το ίδιο ισχύει και για τη λέξη μόνο στην επόμενη παράγραφο. Βλέπω ότι έχει βάλει ερωτηματικό σε αυτό το only, το μόνο η Γιούτα. Αυτά και ίσως επανέρθουμε και καταθέσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για τα σημεία που ανέφερα. Ευχαριστώ Γκέραν ή Ινγκε Γκρέσλε. Υποστηρίζω και εγώ το Ράιμερ Μπέγε. Τα όσα μας παρουσιάζουν ως δίθεν ευκαμψία ε, και να δούμε πού ε, επιτρέψαμε την ευκαμψία, αυτό μας έβγαλε απ' έξω. Όταν τους αφήσαμε να κάνουν αυτοί τις δαπάνες, να αποφασίζουν αυτοί τις δαπάνες, εμείς μείναμε απ' έξω δεν έχουμε λόγο και παρόλα αυτά έχουμε δυσκολίε. Βλέπει για παράδειγμα τον ποινικό αντιδραστήρα του Κοσλοντούι. Ας μην λοιπόν αυτοεξαιρεθούμε εμείς σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού από ε, την διαδικασία που δυστυχώ είναι η γραμμή και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτά δήθεν ως ευκαμψία. Έχω ένα πρόβλημα. έχω μία ερώτηση, γιατί έχω μετά και το θέμα της Λισαβόνας. Την ερώτηση μπορώ να την υποβάλω ήδη, γιατί φοβούμαι να μην χαθεί η ερώτηση. Θέλω να, την, μου απαντηθεί πριν από τις θερινές διακοπές. Μου χρειάζεται ένα λεπτό δηλαδή, για να την υποβάλω. Voilà, mais je ne pas donner... Ναι, αλλά δεν θα μπορέσω να δώσω το, αυτό το λεπτό στην Ίγκε, γιατί ο Υπουργός μόλις ναι, αλλά ούτως ή άλλως ε, είμαι εγγεγραμμένη και στην ε, ε, ημερήσια διάταξη για το θέμα αυτό, γιατί άλλωστε πηγαίνει από κοινού με, την, τη Λισαβόνα. Το σημαντικό είναι να δούμε τι σημαίνει αναδιατύπωση για την Κομισιόν και να ξέρουμε γραπτά από την Επιτροπή ποιες είναι οι δυνατότητες που έχουμε για την αναδιατύπωση, γιατί η δικιά μας νομική υπηρεσία ε, μας προτείνει να ε, ε, να αναφερθούμε σε αυτήν την, και να ζητήσουμε λεπτομέρειες για την αναδιατύπωση. Πολύ ωραία. Ράιμερ, λέει ο πρόεδρος, άκουσες τις απόψεις των συναδέλφων, θέλεις να πεις κάτι, αλλά βεβαίως να σταματήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα γιατί ο καλεσμένος μας είναι ήδη εδώ. Ράιμερ Μπέργκε, ευχαριστώ για την συζήτηση οι λεπτομέρειε ας ρυθμιστούν με τροπολογίες και με συμβαστικές τροπολογίες. Ο Γιώργεν Θάρμ έχει δίκιο ότι με την αλλαγή της διάρθρωσης της έκθεσης μπορεί να οδηγήσει αυτή δηλαδή σε ορισμένες παρανοήσεις με τις νέες διατυπώσεις το θέμα των θετικών και αρνητικών προτεραιοτήτων, το θέμα του τι θεωρούμε εμεί σημαντικό για τον προπολογισμό, πάνω σε αυτά πρέπει να διαπραγματευτούμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αυτά όντω μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιε παρανοήσει. Σωστά το είπε ο κ. Φέρμ. Τα υπόλοιπα όμω θα τα διευκρινίσουμε με τι τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ε, ημερήσια διάταξη. Αναγγέλουμε μονάχα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διατάξεως ότι την 13η Σεπτεμβρίου θα ξανασυνεδριάσουμε. Καλές διακοπές εύχομαι σε όλους και τώρα και κλεισμένο τον...